αγαπητοί συνάδελφοι. Καθίστε παρακαλώ πολύ και ελπίζω να έχετε όλοι τις κάρτες ψηφοφορίας μαζί σας. Ως συνήθως θα κάνουμε πρώτα μια δοκιμαστική ψηφοφορία. άρθη ψηφοφορία. Άρχεται η δοκιμαστική αυτή ψηφοφορία Χρησιμοποιήστε σας παρακαλώ πολύ όλοι τις ε, συσκευές ψηφοφορίας που έχετε μπροστά σας. Ψηφίσατε όλοι στη δοκιμαστική αυτή ψηφοφορία. 35 μέλη, 37 ψήφισαν. Τι, θα γίνει. Α, πολύ ωραία. Λύθηκε το πρόβλημα. Φαίνεται πώς λειτουργούν όλα. Υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση, λίγη ψηφοφορία. Περνάμε τώρα στην πρώτη κανονική ψηφοφορία της ημέρας, στο σημείο 13, προφορική απάντηση για την σύμβαση του Μαυρικίου. Άρχεται η ψηφοφορία. E ένα μέλος του ΕΛΚ παραπάνω Βλέπω ότι ψήφισε. Α, πολύ ωραία. Λύθηκε το πρόβλημα. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με 31 ψήφους υπέρ και 7 αποχές. Περνάμε στο σημείο 14. Ετήσια έκθεση σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Ψηφίζουμε με ανάταση χεριών για την συμβιβαστική τροπολογία 1. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 5. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική τροπολογία 2. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 14. Ψήφι υπέρ. Ψήφι κατά. Αποχές. Νομίζω απορρίπτεται, αλλά α ελέγξουμε ηλεκτρονικά την τροπολογία 14. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 16. Ψήφι υπέρ. Ψήφι κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 17. Υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 19. Υπέρ, κατά, αποχές. Νομίζω πως εγκρίνεται, θα ελέγξουμε όμως καλύτερα ηλεκτρονικά την τροπολογία 19. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 26. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 27. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 28. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Τροπολογία 28. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 34, Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε τώρα για την τροποποιημένη έκθεση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται με 35 ψήφους υπέρ. Συγχαρητήρια. Περνάμε στο σημείο 15. Ο κύριος Μπετίνη θα ήθελε το λόγο. Συγητής, έχει παρακαλώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για την προσπάθεια την οποία κάνανε. Να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της Επιτροπής μας και για τον τριμερή διάλογο και για τον συμβιβασμό στον οποίο καταλήξαμε. Έχουμε θα έλεγα ένα καλό αποτέλεσμα, είναι κάτι το οποίο και το Συμβούλιο θα μπορούσε να αντιμετωπίσει θετικά ε, αναφερθήκαμε και σε σχέση με τις κατεξουσιοδότηση πράξεις και για τα ανθρώπινα δικαιώματα, κάτι που αποτελεί προηγούμενο για μας. Θα σας ευχαριστήσω ε, και όλους τους συνεισηγητές και τις πολιτικές ομάδες. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Μπετίνη. Πράγματι όλη η ομάδα των ε, εισηγητών και των σκιωδών εισηγητών συνεργάστηκε εξαιρετικά και είμαστε με μία ε, φωνή. Και αυτό πραγματικά ήταν ε, πάρα πολύ καλό, είχε εξαιρετικά αποτελέσματα. Το Συμβούλιο συμφώνησε για πρώτη φορά το Κοινοβούλιο να λάβει αυτήν την πράξη κατά εξουσιοδότηση. Είναι λοιπόν μια φωνη και αυτο πραγματικα ηταν παρα πολυ καλο και πολύ το κοινοβουλιο να λαβει αυτην την πραξη κατ' επιτυχία για την Επιτροπή μας αλλά και για το Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ ολόθερμα όλους ε, που συμμετείχατε στην αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου. Έχουμε λοιπόν μπροστά μας το κείμενο και άρχεται η ψηφοφορία. Und Πέρας. 33 ψήφοι υπέρ, 3 κατά, 3 αποχές. Συγχαρητήρια κύριε Σιγητά. Ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι. Σημείο 16. Τίζα. Συμφωνία Τίζα. Τι συναλλαγέ στον τομέα των υπηρεσιών. Να σας υπενθυμίσω ότι στις 9 του μήνα, την επόμενη εβδομάδα, θα διοργανώσουμε ένα ε, χριστουγεννιάτικο ποτό θα λάβετε την πρόσκληση και επίσημα στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο. Θα ήθελα λοιπόν να παρευρεθείτε και να σας ε, ευχαριστήσω όλους για την εξαιρετική δουλειά που κάνατε φέτος. Την επόμενη εβδομάδα λοιπόν. Περνάμε στο σημείο 16. Είναι κάτι που έχουμε συζητήσει ήδη τρεις φορές αυτήν την Επιτροπή. Συμφωνία για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών. 15 Οκτωβρίου ε, έγινε η τελευταία συζήτηση στην Επιτροπή. Μας παρουσίασε η συγγήτρια κυρία Ρέντινγκ την έκθεση. Και στο μεταξύ νομίζω υποβλήθηκαν 599 τροπολογίες. οι οποίες απασχολούν τώρα την εισηγήτρια και τους ε, σκιώδεις εισηγητές και έχουμε γνωμοδοτήσεις από εννέα άλλες επιτροπές. Χαίρομαι λοιπόν πάρα πολύ ε, τώρα που το λόγο θα λάβει η κυρία Ρέντινγκ. Σας ευχαριστώ πολύ αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα να αναφερθώ στα πιο σημαντικά σημεία της έκθεσης αυτής ε, όσον αφορά τις 599 αυτές τροπολογίες τις οποίες έχω λάβει. Λοιπόν, ε, όσον αφορά το πεδίο εφαρμογή των διαπραγματεύσεων. Υπάρχει μια γενικότερη συνένεση στις πολιτικές ομάδες ότι πρέπει να έχουμε συμβατότητα με την Γκάτσα και ότι θα πρέπει να στηρίξουμε το αίτημα της Κίνας να συμμετάσχει και αυτή στις διαπραγματεύσεις. Επίσης, όλοι θέλουν να υπάρχουν διασφαλίσεις όσον αφορά το ανοιχτό διαδίκτυο και την προστασία των κρατών μελών, όσον αφορά τα δικαιώματα των πελατών, των καταναλωτών, Υποστηρίζεται από ό,τι φαίνεται τις προτάσεις μου και μάλιστα επαυξάνεται μέσω περαιτέρω τροπολογιών όσον αφορά το ζήτημα της διαφάνειας. Τα μέλη θέλουν να γίνονται δημόσια τα έγγραφα διαπραγματεύσεων αρκεί να συμμορφώνονται με την πρακτική του ΑΠΟΕ καθώς επίσης και με το κεκτημένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και για όλα τα υπόλοιπα οι περισσότεροι θέλουν να υπάρχει αμοιβαιότητα όσον αφορά ένα κεφάλαιο για τις δημόσιες συμβάσεις και όσον αφορά τον αποκλεισμό των δημοσίων υπηρεσιών. Από ό,τι φαίνεται με τα σημεία αυτά συμφωνούν οι περισσότεροι συνάδελφοι από τις περισσότερες πολιτικές ομάδες. Δεν υπάρχει λόγος να επανέλθουμε στα σημεία αυτά. Είναι τα βασικότερα σημεία συνένεσης και είναι τα βασικότερα σημεία στα πλαίσια διαπραγματεύσεων. Παρ' όλα αυτά κρεμούν κάποια σημεία αμφιλεγόμενα μεταξύ των πολιτικών ομάδων. Πρώτον, όσον αφορά την πρόσβαση στι αγορέ. Ορισμένοι ευρωβουλευτές θέλουν ε, ιδιαίτερα φιλόδοξες δεσμευσεις στον τρόπο 1 και 4, ενώ άλλα μέλη είναι κατά των περαιτέρων δεσμεύσεων πέρα από τον ΚΑΤΣ, όσον αφορά το MODE 1 και το MODE 4. Και ορισμένοι ευρωβουλευτές θέλουν διατηρήσουμε το εφιστάμενο πλαίσιο των πραγματεύσεων, ενώ πάλι άλλοι αντιτίθενται σε οποιοσδήποτε ρήτρες διατήρηση τη ισχύω κατάσταση ή ρήτρε προσαρμογής. Πιστεύω όμω ότι για τα σημεία αυτά που υπάρχει διαφωνία θα καταφέρουμε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία. Όσον αφορά τον τρόπο 4, το ΜΟ 4 πιο συγκεκριμένα, που έχει να κάνει με την προσωρινή κινητικότητα των υψηλά εξειδικευμένων επαγγελματιών. Έχουμε εδώ πέρα πολλέ τροπολογίε και υπάρχει ένα έντονο ενδιαφέρον. Αναφερόμαστε εδώ πέρα όμω και στη σύμβαση του ILO, καθώ επίση και στη νέα οδηγία τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την απόσπαση των εργαζομένων και γίνεται επίση και μία αναφορά στι δοκιμέ οικονομικών αναγκών των κρατών μελών. Και για το σημείο μα αυτό πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να καταλήξουμε σε συνένεση. Όσον αφορά τώρα την εγχώρια νομοθεσία, ορισμένε πολιτικέ ομάδε είναι λίγο πιο επιφυλακτικέ όσον αφορά τα λεγόμενα necessity tests, δοκιμές αναγκαιότητος. Από ό,τι φαίνεται όμως οι περισσότεροι θεωρούν ότι δεν θα πρέπει να προβλέπετε εδώ πέρα τίποτα πιο περιοριστικό από ό,τι ήδη προβλέπεται στα πλαίσια της GATS και από ό,τι ήδη ισχύει στο νοσιακό δίκαιο. Κύριε Πρόεδρε, λοιπόν, είναι σαφές ότι υπάρχει ένα μεγάλο περιθώριο για να καταλήξουμε σε συμβαστικές προτάσεις και ως εισηγήτρια είμαι σε επαφή με τους συνεργάτες μου και απευθύνομαι σε όλες τις πολιτικές ομάδες προκειμένου να καταλήξουμε στις καλύτερες δυνατές συμβαστικές λύσεις. Και βλέπετε ότι η ίδια η αρχική μου έκθεση είχε μια συμβαστική φύση, αλλά βέβαια μπορούμε να πετύχουμε ακόμα περισσότερους συμβασμούς. Σε συνεργασία λοιπόν με τους κοιόδης ε, εισηγητές θα έχουμε μια πολύ θετική συνεργασία πιστεύω και ήδη να τους ευχαριστήσω για την πολύ φιλική και επικοδομητική στάση που είχαν στα πλαίσια των προηγούμενων συζητήσεων. Θα λάβουμε υπόψη μας ε, τις περισσότερες προτάσεις που έχουν κάνει οι συνάδελφοι από την Επιτροπή ΙΝΤΑ, ενώ θα προσπαθήσουμε να συντάξουμε τις συμβαστικές τροπολογίες και θα προσπαθήσω να συμπεριλάβω επίσης και τις ε, απόψεις των υπόλοιπων επιτροπών που γνωμοδοτούν και δεδομένου ότι είναι ιδιαίτερα ευρύ το φάσμα των διαπραγματεύσεων αυτών, οι δικοί μας, μάλλον οι προτάσεις των υπολείπων επιτροπών είναι πάρα πολύ σημαντικές. Γι' αυτό το λόγο προσπαθούμε επί του παρόντος να αφομοιώσουμε, να συμπεριλάβουμε στην πρότασή μας τις περισσότερες γνωμοδοτήσεις των υπολείπων επιτροπών. Ένα χρόνο λοιπόν μετά την παρακολούθηση κάθε σταδίου των διαπραγματεύσεων αυτών, βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανταποκρίθηκε στα δικά μας θετήματα. Ερχόταν δηλαδή στο Monitoring Group, στην ομάδα αυτή παρακολούθησης, έδινε εξηγήσει σε αντίθεση με ό,τι έγινε στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης. Εμείς στην ομάδα monitoring, στην ομάδα παρακολούθησης, είχαμε πολύ καλή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υψηλότατο επίπεδο διαφάνειας και ως Ευρωβουλευτές θα πρέπει να θέσουμε σαφείς κατευθύνσεις για το τι θέλουμε να πετύχουμε και τι θέλουμε να αποφύγουμε. Αυτός είναι ο απότερος στόχος άλλωστε και του ψηφίσματος αυτού. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο χρειαζόμαστε μια πολύ σημαντική πλειοψηφία τόσο στην Επιτροπή μας όσο και στην Ολομέλεια. Αν ο πραγματικός μας στόχος είναι να πούμε ξεκάθαρα προς τις διαπραγματευτές, κοιτάξτε, αυτά θέλουν οι εκπρόσωποι των Ευρωπαίων πολιτών. Αυτά θέλουν να συμπεριληφθούν στην ΤΙΖΑ. Τότε αυτό δεν μπορούμε να το πετύχουμε μια μικρή ασθενή πλειοψηφία στην Ολομέλεια. Χρειαζόμαστε ισχυρή πλειοψηφία. Δεν θα ψηφίσουμε λοιπόν την ίδια τη συμφωνία ΤΙΖΑ. Θα ψηφίσουμε υπέρ ή κατά μια συμφωνία πριν την ολοκλήρωση τη συμφωνία αυτή. Ουσιαστικά προσπαθούμε εμεί να δώσουμε συστάσει αυτή τη στιγμή κατευθύνσει προ του αρμόδιου διαπραγματευτέ. Και όλε οι πολιτικέ ομάδε και ευρωβουλευτέ που θέλουν τη συμφωνία αυτή θέλουν η συμφωνία αυτή να λειτουργεί υπέρ των επιχειρήσεων και υπέρ των πολιτών μα. Δεν πρέπει λοιπόν να χάσουμε τη σημαντική αυτή ευκαιρία που μα δίνεται αυτή τη στιγμή. Και προφανώ είμαι ακόμα και σήμερα στη διάθεσή σα για να ακούσω τι παρατηρήσει σα και να συνεχίσουμε τον πολύ αυτοεπικοδομητικό διάλογο που έχουμε ήδη ξεκινήσει μεταξύ των πολιτικών ομάδων και είναι πολύ σημαντικό να διατηρήσουμε την εξαιρετική αυτή συνεργασία που ήδη έχω με τους σκιώδες συγητές. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Ρέντιν. Πολλά υποσχόμενη ήταν η παρουσίασή σας. Είναι πολύ ευχάριστο το ότι καταφέρατε να συμφωνήσετε για αυτά τα τέσσερα σημεία με τους σκιώδες εισηγητές και σας συγχαίρω γι' αυτό. Θα δώσω τώρα στην κυρία Κέρτον Ντάρλινγκ και ο διεξηγήτρια το λόγο. Παρακαλώ. Οι διαπραγματεύσει τη πράγματι προκαλούν όλο και περισσότερη προσοχή και εντό και εκτός κοινοβουλίου. Νομίζω ότι ένα από τα βασικά συμπεράσματα που βγαίνει από το συγκεκριμένο ψήφισμα είναι ο τρόπος με τον οποίο σαν Κοινοβουλευτική Επιτροπή συνεργαστήκαμε με τις άλλες επιτροπές που εκφέρουν γνωμοδοτήσεις για να διαμορφώσουμε τη θέση του Κοινοβουλίου. Θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν τον εισηγητή για τη δεκτικότητά του και τη διαφάνεια της δουλειάς του μέχρι τώρα. Πολλές τοπολογίες και από εμά και από τις νομοδότριες κοινοβουλευτικές επιτροπές. Είμαστε στο μέσο της διαδικασίας, στην παρούσα φάση, σκεφτόμενος τι πιθανές ε, συμβιβαστικές προτάσεις έχουμε. Αυτό δείχνει όμως ότι υπάρχει μια ηγετική θέση του Κοινοβουλίου ε, σε σχέση με τα σχόλια τα οποία απαιτούν γενικότερα στον κόσμο μεγαλύτερη διαφάνεια στις εμπορικές διαπραγματεύσεις. Εμείς δεν μπορούμε άμεσα να ελέγξουμε φυσικά τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η διαπραγματευτική ομάδα στην ε, διαπραγμάτευση. Παρ' όλα αυτά απαιτούμε να υπάρχει ένα υψηλό επίπεδο διαφάνειας και δεκτικότητας. Να διευκρινίσω προς την κυρία Ρέντινγκ ότι το ψήφισμα αυτό δεν είναι υπέρ της αποδοχής ή της απόρριψης μιας εμπορικής συμφωνίας που δεν υπάρχει ακόμα. Το θέμα είναι να μπορέσουμε να επηρεάσουμε τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις και ο καλύτερος τρόπος που θα μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό είναι να προσδώσουμε μεγαλύτερη διαφάνεια στη συζήτηση για το κλίμα και να χρησιμοποιήσουμε το ψήφισμα αυτό για να δείξουμε ακριβώς τι θέλουμε να υπάρχει και τι δεν θέλουμε να υπάρχει σε ένα κάποιο τελικό κείμενο. Έχουμε πολλές τοπολογίες καταθέσει για να παρουσιάσουμε τις θέσεις μας. Το κομβικό σημείο θα έλεγα είναι η συνεκτικότητα. Εμείς το συζητήσαμε, μάλλον συζητήσαμε το θέμα του TTIP και γι' αυτό πρέπει να υπάρχει συνοχή με τις προτάσεις που έχουμε ε, ήδη δεχτεί σε σχέση με το TTIP. Η TISA είναι μια καλή θα έλεγα ευκαιρία για να κλείσουμε τα κενά και να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις ε, του διαδικτύου. Έχουμε όμως διευκρινίσει σαφώς ότι οι δημόσιες υπηρεσίες μας, οι συνθήκες εργασίας επίσης, δεν είναι υποσυζήτηση και δεν θα πρέπει να επηρεαστούν αρνητικά από την ΤΙΣΑ. Θέλουμε εμείς να επιβεβαιώσουμε το δικαίωμα των δημοσίων αρχών να διακανονίζουν, να ορίζουν τις συνθήκες εργασίας και τις αντίστοιχες ρήτρες. Αυτό είναι κάτι το οποίο απαιτεί λίγο περισσότερο από μία απλή αναφορά σε σχέση με την προστασία των προσωπικών δεδομένων επίσης είναι θέμα το οποίο θα πρέπει με τις συμβιβαστικές τροπολογίες να καλυφθεί και πηγαίνουμε προς την κατεύθυνση αυτή και το θέμα με την TISA και την TIP φυσικά είναι ότι είναι μια καλή ευκαιρία να προωθήσουμε τον πολυμερή τρόπο θα έλεγα συνεργασία σε οικονομικό και εμπορικό επίπεδο με τον υπόλοιπο κόσμο στον κόσμο. Να μην υπάρχουν μόνο διμερείς σχέσεις ανάμεσα στις μεγάλες πλούσιες χώρες, αλλά να υπάρξει μια συμφωνία ωφέλιμη για όλες τις χώρες του κόσμου και να αντιμετωπιστεί και το θέμα ε, των, ε, παρα... των κλεψιτήπων προϊόντων όπως και του κοινωνικού ντάμπινγκ στην Ευρώπη. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει λοιπόν ό,τι μπορεί έτσι ώστε το ΤΙΣΑ να είναι μια πολυμερή συμφωνία και ε, να ε, μην υπάρχουν ε, ρυθμίσεις οι οποίες να είναι διαφορετικές από τις συνθήκες, από τις ρήτρες, our work, uh, in our first... από τις ρήτρες γάτ. Είχαμε μια πρώτη συνάντηση των σκιωδών, θα υπάρξει και άλλη μια στο τέλος της εβδομάδας Νομίζω ότι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε μια καλή θα έλεγα πορεία και να καλύψουμε τις ανησυχίες όλων των συναδέλφων. Περιμένω από τον εισηγητή να είναι ακόμα πιο δεκτικός στις συμβιβαστικές προτάσεις στο μέλλον. Ευχαριστώ Πρόεδρε, να ευχαριστήσω την εισηγήτρια. Χαίρομαι πάρα πολύ για την ιδιαίτερη επικοδομητική εργασία που έχει κάνει η εισηγήτρια καθ' όλη τη διάρκεια αυτή τη διαδικασία. Είχαμε μια πολύ θετική συνεργασία, όπω είπε και η εισηγήτρια, με όλου του κοιόδη εισηγητέ. Προσπαθούμε να συμπεριλάβουμε όλε τι διαφορετικέ απόψει, όλε τι διαφορετικέ ερμηνείε για το τι μπορούμε να πετύχουμε στα πλαίσια της συμφωνίας αυτής για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών και ελπίζω ότι θα καταφέρουμε να διευθετήσουμε όλα τα προβλήματα μέσω των συμβαστικών τροπολογιών. Είχαμε σημειώσει πρόοδο στις πρώτες συνεδριάσεις των σχεδόν εισηγητών και ευελπιστώ ότι θα καταφέρουμε να καταλήξουμε σε θετικά αποτελέσματα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε ενδεχομένω τα βασικότερα ζητήματα τα οποία μας αποσχίλησαν στην πρώτη συνεδρίαση των σχεδόν εισηγητών. Από την πρώτη λοιπόν συζήτηση που είχαμε, βλέπουμε ότι η ρήτρα διατήρηση τη ισχύουσας κατάσταση και η ρήτρα προσαρμογή θα αποτελέσουν μήλον τη έρηδο κατά τη διάρκεια των συζητήσεων. Εγώ θεωρώ ότι οι δύο αυτές ρήτρες διατήρησης ισχύουσας κατάστασης και ρήτρα προσαρμογής θα πρέπει να διατηρηθούν προκειμένου να μην υπάρχει κατάχρηση των διατάξεων της συμφωνίας αυτής από τις τρίτες χώρες κάθε φορά που θέλουν να παρέχουν συγκεκριμένες υπηρεσίες, κυρίως δημόσιας φύσης, στα κράτη-μέλη. Όσον αφορά το θετικό και αρνητικό κατάλογο, το μοντέλο το οποίο προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι το θετικότερο, δίνει μια κάποια ευελιξία και από την άλλη ένα κάποιο έλεγχο όσον αφορά την πρόσβαση στις αγορές. Πολλές φορές βλέπουμε ότι υπάρχουν ε, ορισμένοι οι οποίοι δεν συμμερίζονται το ίδιο επίπεδο φιλοδοξίας ε, στα πλαίσια αυτής της συμφωνίας. Για να είμαι λίγο πιο συγκεκριμένοι, θα μπορούσαμε να αφαιρθούμε σε κάποιες συγκεκριμένες τροπολογίες, την υπαριθμών 23 και 32, που αναφέρονται στην πρόσβαση στις αγορές. Θα ήθελα να τονίσω τις συζητήσεις που ήδη έχουμε όσον αφορά τις τροπολογίες εκείνες που αναφέρονται στον αποκλεισμό των οπτικοακουστικών και πολιτιστικών υπηρεσιών. Μπορώ να συμφωνώ με την οπτικοακουστική εξαίρεση εφόσον υπάρχει συγκεκριμένο ορισμός. Από την άλλη έχω κάποιες ενστάσεις όσον αφορά την εξαίρεση η οποία προτείνεται για τις πολιτιστικές υπηρεσίες για τις οποίες δεν υπάρχει συγκεκριμένο ορισμός. Νομίζω ότι η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα επιθετικό συμφέρον στο ζήτημα αυτό όσον αφορά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τις διαφημίσεις και νομίζω ότι αυτό μπορεί ενδεχομένως να αποδυναμωθεί αν έχουμε έναν γενικό και αόριστο αποκλεισμό όσον αφορά τις πολιτιστικές υπηρεσίες. Ξέρετε ότι και σε σχέση με, το, με τη συμφωνία TTIP νομίζω ότι θα πρέπει να ακολουθήσουμε την τροπολογία 23 αλλά διατηρήσουμε παράλληλα και τα όσα λέγονται στην τροπολογία 32 όσον αφορά την διατήρηση της γλωσσικής πολυμορφίας. Να αναφερθώ και σε κάτι ακόμα το οποίο μου απασχολεί ιδιαίτερα και το οποίο αντιτίθεται στην γενικότερη ιδέα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, ευρωπαϊκή πράξη επιχειρήσεων. Όντως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν πέτυχε τον κατάλληλο βαθμό αμοιβαιότητος με τις τρίτες χώρες όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις. Το είχαμε πει ήδη αυτό και στο παρελθόν και αργότερα σήμερα θα μας απασχολήσει και το ζήτημα αυτό με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ποια θα είναι τα επόμενα βήματα. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι λανθασμένο να συμπεριλάβουμε το European Business Act στα πλαίσια της ΤΙΖΑ, γιατί δεν έχει αποσαφηθεί ακόμα η δική μας στάση σε σχέση με τις δημόσιες συμβάσεις και την πράξη αυτή. Τέλος, εφόσον μιλάμε για την αμοιβαιότητα, το ζήτημα αυτό προκύπτει με κάποιες επιμέρους τροπολογίες. Συμφωνώ με την εισηγήτρια ότι το ζήτημα αυτό θα πρέπει να μας απασχολήσει και θα πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί. Από την άλλη αποτελεί ένα τμήμα επιθετικής πολιτικής της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γίνεται μια κλίση για μηδεότητα, αλλά από την άλλη βλέπουμε ότι οι δεσμεύσεις των τρίτων χωρών δεν είναι όσο φιλόδοξες είναι οι δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι μέσω της συμφωνίας αυτής θα πρέπει να ανεβάζουμε τον πύχη και όχι να ψάχνουμε τον ελάχιστο κοινό παρανομαστή. Είναι πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να καταλήξουμε σε ένα ψήφισμα το οποίο θα είναι σαφές, θα έχει μια συγκεκριμένη αποφασιστικότητα για να καταλήξει σε μια καλή εμπορική πολιτική, σε μια καλή εμπορική συμφωνία. Μια τίζα που θα λειτουργεί υπέρ των πολιτών μας. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι και θα πρέπει να δώσουμε έναν αγώνα για να πετύχουμε μια πολύ καλή συμφωνία. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν το μήνυμα που θα στείλει η Επιτροπή μα και γενικότερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ότι θέλουμε να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στα πλαίσια τη ΤΙΖΑ μάλιστα, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Οι συναδελφοί είπαν πάρα πολλά, οπότε θα είμαι σύντομη. Καταρχάς εκτιμώ την συλλογή ε, πληροφοριών της εισηγήτριας και εκτιμώ πάρα πολύ το γεγονός ότι προσπάθησε να βρει μια συνένεση ανάμεσα στους σκιώδεις εισηγητές. Είμαι πεπισμένη ότι θα καταφέρουμε να στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα στους διαπραγματευτές. Δεν πρόκειται για την τελική κρίση αυτή τη στιγμή. Θα ήθελα λοιπόν να παροτρύνω όλους ε, όσοι ε, εμπλέκονται με το θέμα αυτό να εστιάσουν στα ουσιώδη παρά ε, να γενικεύουν παρά να ασχολούνται με πολλά τα οποία θα αποδυναμώσουν το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε και θα αποδυναμώσουν και την ευκαιρία που ε, έχουμε να κατευθύνουμε τις διαπραγματεύσεις σε ένα καλό αποτέλεσμα. Πολλά διακυβεύονται αυτή τη στιγμή, οι υπηρεσίες γίνονται λένε και σημαντικότερες στην παγκόσμια οικονομία και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια αρκετά ανοιχτή αγορά. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω πως ε, είναι μια πάρα πολύ σημαντική ευκαιρία να γίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση πιο ανοιχτή. Δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα, αντιθέτως έχουμε να κερδίσουμε πάρα πολλά. Έχουμε πάρα πολύ καλά καταρτισμένο ε, εργατικό δυναμικό το οποίο θα μπορούσε να μας ωφελήσει. Επίσης, ας μην ξεχνάμε πως ε, μπορούμε να ενισχύσουμε και να ανεβάσουμε τα παγκόσμια πρότυπα και να ανεβάσουμε τον πύχη σχετικά με τους ε, κανόνες ε, της ε, αγοράς. Η πρόσβαση στην αγορά είναι πάρα πολύ σημαντική. Εξίσου σημαντικά όμως είναι και τα επόμενα βήματα. Μια πολυμερή συμφωνία θα είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό μήνυμα. Και πιστεύω πως πρέπει να στείλουμε το μήνυμα πως επιθυμούμε να συμπεριληφθούν και άλλες χώρες, οι χώρες BRICS, η Κίνα, και άλλες ώρες ε, στις, ε, στο εμπόριο υπηρεσιών. Οι ψηφιακές υπηρεσίες επίσης γίνονται όλο ένα και πιο σημαντικές. Γι' αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό να δημιουργηθούν οι κατάλληλοι κανόνες. Εμείς θα θέλαμε να ε, επικαιροποιηθεί η ΓΚΑΤ στα πλαίσια της συμφωνίας ΤΙΣΑ από τη μία για να διασφαλίσει την ελεύθερη ροή των πληροφοριών και από την άλλη φυσικά να γίνονται, να γίνονται σεβαστοί τα προσωπικά δεδομένα και τα ατομικά δικαιώματα των ε, πολιτών. Θα θέλαμε λοιπόν η συμφωνία να είναι φιλόδοξη. Πιστεύουμε πως είναι σαφώς ε, ε, στο συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι φιλόδοξη η συμφωνία. Προσβλέπουμε στην διαφάνεια και στην καθολική πρόσβαση όλων των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο κείμενο. Και η ομάδα μου και εγώ πιστεύουμε ότι η διάθεση περισσότερων πληροφοριών στο κοινό θα συνεισφέρει σε μια καλύτερη ανταλλαγή απόψεων και θα μας επιτρέψει να ε, με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς οι οποίοι επίσης έχουν πολύ ψηλέ απαιτήσει. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε ένα πρόβλημα με το χρόνο. Στις 11 θα έρθει ο Υπουργός του ε, Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και πρέπει να έχουμε τελειώσει μέχρι ε, τότε. Διαφορά θα πρέπει να διακόψουμε τη συζήτηση και να αρχίσουμε στις 11.45. Ο κύριος Κούλογλου έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είμαι σκιώδης εισηγήτρια για τη δική μας πολιτική ομάδα. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Ρέντινγκ για την προσπάθεια την οποία έκανε για την έκθεση αυτή θέλουμε να υπάρξει μια τέτοια συμφωνία, αλλά δεν θα πρέπει να είναι εις βάρος του κοινού καλού και των πολιτών της Ένωσης. Οι ανησυχίες μας δεν έχουν ακόμα διαλυθεί για τη μεγαλύτερη διαφάνεια. Το έχει ήδη ζητήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα αποτελέσματα μέχρι τώρα είναι ανεπαρκή. Η κοινωνία των πολιτών, οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις και τα συνδικάτα αντιμετωπίζουν τα ίδια εμπόδια με το παρελθόν ε, για ενημέρωση και έχουν πάντα πάρα πολλές ανησυχίες. Εμείς θα θέλαμε να υπάρξει πλήρης σεβασμός των δικαιωμάτων μας σε σχέση με τον έλεγχο της συγκεκριμένης αυτής συμφωνίας. Θέλουμε ένα κεφάλαιο που να περιλαμβάνει τις βασικές αρχές του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας. Αυτό το κεφάλαιο θα πρέπει να είναι δεσμευτικό για όλους τους υπογράφοντες. Θα πρέπει επίσης να υπάρξει απόρριψη των ε, ρητρών, ε, το να υπάρξει απόρριψη αυτών των ρητρών που έχουν ήδη ονοματιστεί όπως τα standstill δεν αρκεί. Δεν θα πρέπει να διευκρινίζεται ότι δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα στο σύνολο της έκθεσης. Γιατί υπάρχουν πολλοί οι οποίοι προωθούν από τη μία τα πλεονεκτήματα των πολυμερών σχέσεων και από την άλλη δίδουν τον ε, ρόλο της χώρας παρατηρητή σε οποιαδήποτε χώρα το επιθυμεί. Νομίζουμε επίσης ότι ο αρνητικός κατάλογος ε, είναι κάτι το οποίο μπορεί να αποτελέσει απειλή για τα δικαιώματά μας στον τομέα τον περιβαλλοντικό, τον παραγωγικό και τον ε, εργασιακό. Σκα. Ευχαριστώ την εισηγήτρια, ευχαριστώ και τους σκιώδεις εισηγητές. Έχω κάποια θέματα που θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικά. Το θέμα του πολυμερούς χαρακτηριστικού είναι σαφές η ΤΙΖΑ να λειτουργήσει σε αυτό το επίπεδο. Υπάρχουν ορισμένες τροπολογίες οι οποίες ξεπερνούν τα γκάτ και νομίζω ότι δεν είναι δυνατόν με τον τρόπο αυτό να πετύχουμε το στόχο που έχουμε και αυτό μας ανησυχεί. Η ιδέα αυτή των πολυμερών σχέσεων θα πρέπει να χαρακτηρίζει όχι μόνο την ΤΙΖΑ αλλά και όλα τα παραρτήματα. Και δεν μπορούμε να δεχθούμε προτάσεις σχετικές με τις ρήτρες αυτές της Standstill θα πρέπει να εμείνουμε επίσης σε σχέση ε, με, τις, ε, με τους θετικούς καταλόγους για την ελεύθερη πρόσβαση. Τώρα για τις δημόσιες προμήθειες, ε, εδώ μπορεί να υπάρχουν στοιχεία που είναι αντίθετα με τον πολυμερή χαρακτήρα και ξέρουμε ότι ο ΠΟΕ λειτουργεί ουσιαστικά ιδιαίτερα με διμερεί σχέσει και αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα σε πολλές χώρες. Οπότε θα πρέπει να υπάρχει μια ρήτρα opt-in, μια ρήτρα συμπερίληψη για τις χώρες που το επιθυμούν. Ε, οι εθνικές ρυθμίσεις είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Πρέπει να υπάρχει μια ρήτρα η οποία λέει ότι το δικαίωμα των νομοθετικών ρυθμίσεων σε εθνικό επίπεδο θα πρέπει να διασφαλιστεί νομικά. Και ταυτόχρονα λέμε ότι για να είμαστε συνεκτικοί με την αρχή της πολυμέρειας τότε θα πρέπει τα θέματα τα οποία ακαλύπτονται από το άρθρο 6 της Συμφωνίας ΓΚΑΤ σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει σώνη και καλά ένα τεστ αναγκαιότητας, ένας έλεγχος αναγκαιότητας των προτινόμενων ρυθμίσεων. Όλα αυτά θα πρέπει να είναι συμβατά βέβαια και με το ισχύον και το μελλοντικό πλαίσιο σεβασμού των προσωπικών και εμπιστευτικών δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον υπόλοιπο κόσμο. Και για άλλους τομείς πρέπει να υπάρχει αυτή η συνεκτικότητα θα πρέπει επίσης να είμαστε συνεκτικοί και με την γνωμοδότηση που ήδη ψηφίστηκε και κυκλοφόρησε από πλευράς της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων. Οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες είναι ένα προβληματικό για μας θέμα. Πρώτα θα πρέπει να δούμε τα αποτελέσματα των προηγούμενων ρυθμίσεων και σε ποιο βαθμό ε, επηρέασαν την κρίση και το θέμα της πρόσβασης στις αγορές θα πρέπει να υπάρχει ένας έλεγχος εκ των προτέρων για τον τομέα αυτό. Και για τις δημόσιες υπηρεσίες δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, γνωρίζετε τις απόψεις μας πάνω σε αυτό. Θα συμφωνήσω και με το SND. Θέλουμε να, έχουμε πάντα υπόψη στις ρυθμίσεις και τις αναπτυσσόμενες χώρες. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την συνάδελφο Ρέντινγκ για την εξαιρετική της συνεργασία με τους κοιόδης ηγητές προκειμένου να καταλήξουμε σε μια συμβαστική λύση. Εμείς είμαστε κατά της βασικής αρχής όσον αφορά αυτές τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών, θεωρούμε πάντως ότι θα πρέπει να υπάρχουν καταχρήσεις. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι υπάρχει μια μυστικότητα όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις για την ΤΙΖΑ. Αυτό ανησυχεί και εμάς και τους πολίτες. Γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι η δική μας έκθεση αποτελεί ευκαιρία προκειμένου να καθησυχάσουμε τους πολίτες και να επιθυμίσουμε στις διαπραγματευτές για ποια σημεία εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε πίσω. Εμείς ως Ευρωβουλευτές δεν θα πρέπει να εθελοτυφλούμε αυτή τη στιγμή για το πώς έχει πραγματικά η κατάσταση. Δεν μπορούμε με κλειστά μάτια να αποδεχθούμε τα όσα αποφασίζονται και κλεισμένων των θυρών. ευχαριστήσω λοιπόν τη συνάδελφο Ρέντινγκ για την έκθεσή της. Το αρχικό της κείμενο ήταν πολύ καλύτερο πάντως από αυτό το οποίο βλέπουμε στις τελευταίες συνεδριάσεις. Δεν είμαι ικανοποιημένη με την τροπή που παίρνει η έκθεση αυτή όπως και για το ψήφισμα για το τύπη, φαίνεται ότι οι πολιτικές ομάδες πιέζουν προς μια γενική συμφωνία η οποία θα καλύπτει τους πάντες αλλά δεν θα εμβαθύνει σε καθόλου λεπτομέρειες πιστεύω ότι οι πολίτες χρειάζονται κάτι πολύ καλύτερο, όχι ένα γενικό κείμενο το οποίο δεν θα προβλέπει συγκεκριμένες διασφαλίσεις κατά της απελευθέρωσης των υπηρεσιών. Ορισμένοι συνάδελφοι θέλουν να συμπεριλάβουν κάποια ευαίσθητα ζητήματα στην έκθεση αυτή όπως ένα θετικό κατάλογος για τις δημόσιες υπηρεσίες ή αποκλεισμό των υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος, καθώς επίσης και το ζήτημα του domestic regulation, των χώριων νομοθεσιών. Αν εμείς δεν αναλάβουμε αυτή την αρμοδιότητα να θέσουμε συγκεκριμένε διασφαλίσεις, πραγματικά ποιος πρόκειται να το κάνει στη θέση μας. Χρειαζόμαστε ένα νέο κείμενο, όχι ένα κείμενο το οποίο θα είναι πανομοιότυπο με αυτό τη TTIP. Θέλουμε πραγματικά να καταφέρουμε να επηρεάσουμε τις διαπραγματεύσεις. Νομίζω ότι θα πρέπει να χάσουμε την καταπληκτική αυτή ευκαιρία που μα δίνεται. Σα Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Από ό,τι φαίνεται η έκθεση αυτή ακολουθεί το δρόμο της έκθεσης που συντάξαμε για το TTIP. Ξεκινάμε πολλές καλές θετικές προθέσεις, αλλά στο δρόμο βλέπουμε ότι καταλήγουμε απλώς σε έναν κατάλογο θετικών προθέσεων με κίτρινες και κόκκινες γραμμές που πολύ φοβάμαι τελικά ότι δεν θα σεβαστεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τι μπορούμε λοιπόν εμείς να κάνουμε σε σχέση με όλα αυτά λέγεται σε ένα σημείο ότι ένα από τα κεφάλαια της TTIP αφορά το πετρέλαιο και ότι συντάχθηκε μαζί με τους εκπροσώπους του κλάδου του πετρελαϊκού θα συμβεί κάτι τέτοιο και στην Τίζα. Ξέρετε ότι τα δύο τρίτα του ΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιστοιχούν στις υπηρεσίες. Νομίζω λοιπόν ότι δεν θα πρέπει το ζήτημα αυτό να βγει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης κατά αυτόν τον τρόπο. Νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει μια απόλυτη διαφάνεια για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Δεν έχω να πω ακόμα πάρα πολλά πράγματα επί της ουσίας. Αυτό το οποίο βλέπω πάντως είναι ότι έχουμε μπροστά μας μια επικείμενη συμφωνία που αναφέρεται σε παγκόσμια πρότυπα, προσπαθεί να διατηρήσει το δικαίωμα της εγχώριας νομοθεσίας Υπάρχουν όμω πάρα πολλά σημεία τα οποία δεν έχουν διευθετηθεί και γενικά θα είναι πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί αυτή η συμφωνία. Η ΤΙΖΑ θα έχει και ένα κεφάλαιο για την εγχώρια νομοθεσία, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι η ίδια αυτή η συμφωνία θα επηρεάσει τον τρόπο χάραξη εθνική πολιτική. Επομένω, προβλέπετε όπω και για το TTIP ένα διαιτητικό δικαστήριο και για την ΤΙΖΑ. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα για ένα λεπτό ο κύριο και ο κύριο Χέλνερ. Ναι κύριε Πρόεδρε, πράγματι έχει υπάρξει μια πολύ σημαντική προσπάθεια από τους εισηγητές, από την εισηγήτρια και τους κοιόδης εισηγητές καλύτερα. Αυτό νομίζω ότι αντακατοπτρίζει και την, το ενδιαφέρον ενός μεγάλου αριθμού των συμπολιτών μας και μια ανησυχία που έχουν η οποία είναι απόλυτα νόμιμη θα έλεγα και δεν μπορούμε να απαντήσουμε μέσω παιδαγωγικών ρυθμίσεων που λέγουν ότι απαιτείται ε, μέγιστη δυνατή διαφάνεια και έτσι όλα θα πάνε καλά. Το θέμα δεν είναι μόνο παιδαγωγικό, το θέμα είναι να γνωρίζουν οι πολίτες τι σημαίνουν τα αποτελέσματα των φιλευθεροποιήσεων στον υπόλοιπο κόσμο. Και ακριβώς εδώ τίθεται το θέμα ε, της ε, σωστής ή μη της ορθότητας ή μη αυτής της διαπραγματευση μιας τέτοιας διαπραγμάτευσης. Γιατί θα μπορούσαμε να καλύψουμε τις ανάγκες στον ψηφιακό τομέα και όχι να συμπεριλάβουμε πάρα πολύ περισσότερους τομείς και υπηρεσίες. Υπάρχει ένα ψήφισμα του Κοινοβουλίου το 2013. Έλεγε το ψήφισμα αυτό. Δεν θα πρέπει να συμπεριληφθούν οι πολιτιστικές υπηρεσίες, όλοι το υπερψήφισαν αυτό και η δεξιά έπρεπε να υπάρχουν μόνο θετικοί κατάλογοι και το υπεψήφισε και η δεξιά και αυτό το οποίο έχει σημασία είναι ότι δεν μπορεί να υπάρξει ρήτρα status quo και ρήτρα standstill γιατί αυτό σε επίπεδο δημοκρατίας δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα. Κύριε Φιάινερ, ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι σύντομο. Καταρχά, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον, την εισηγήτρια και του σκιώδει εισηγητέ και θα ήθελα να πω τα εξή ε, σύντομα. Καταρχάς, πρέπει να στοχεύουμε στο να δημιουργήσουμε ένα φιλόδοξο, άρκετα φιλόδοξο κείμενο. Αυτός είναι ένας ε, τομέας όπου φαίνονται ξεκάθαρα τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην δημιουργήσουμε νέε κόκκινες ε, γραμμέ. Διότι αν κοιτάξουμε το, την παγκόσμια κατάσταση στο εμπόριο υπηρεσιών θα δούμε την θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν πρέπει να ε, είμαστε ε, λοιπόν αμυντικοί. Πρέπει να έχουμε σαφείς στόχους. Έπειτα, η ροή των δεδομένων. Η μεταφορά δεδομένων είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα στις ε, ψηφιακές υπηρεσίες. Και είναι πάρα πολύ ε, σημαντικό για μεταποιητικό τομέα. Πρέπει να συνδυαστεί όμως και με την ε, κατανόηση αυτής ε, της ροής δεδομένων, διότι δεν μπορούμε να έχουμε ελεύθερη ροή δεδομένων χωρίς προστασία δεδομένων ή προστασία δεδομένων χωρίς ε, ροή δεδομένων. Πρέπει λοιπόν να το προσέξουμε αυτό και να καταφέρουμε να συνδυάσουμε και τα δύο. Και τέλος, σχετικά με τις οπτικοακουστικές υπηρεσίες, αναγνωρίζω ότι είναι ένα ευαίσθητο θέμα για αρκετούς, γι' αυτό χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Και εδώ συμφωνώ με την ΕΜΑ και πιστεύω πως πρέπει να είμαστε απόλυτα σαφείς στο τι επιθυμούμε. Και να μην ε, αναλωνόμαστε με το τι δεν είναι σωστό και το τι είναι λάθος, αλλά με το τι θέλουμε. Πρέπει να, να χρησιμοποιήσουμε επίσης τις εξαιρέσεις που έχουμε στη διάθεσή μας, παρά να βγάζουμε ολόκληρα μπλοκ ε, από τις διαπραγματεύσεις. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να κρατήσουμε το δικαίωμα που έχουμε να κάνουμε εξαιρέσεις. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ σύντομα κύριε Πρόεδρε. Ακούσαμε τα σημαντικότερα σημεία. Θα πρέπει απλώς να συντοπίσουμε εδώ πέρα ότι πρέπει να πετύχουμε μια συμφωνία στις διάφορες πολιτικές ομάδες. Υπήρχε μεγάλη απόκληση απόψεων στην αρχή, αλλά τώρα από ό,τι φαίνεται συμφωνούμε ότι η συμφωνία ΤΙΖΑ μπορεί να μειώσει τη φτώχεια και τις ανισότητες και ότι μπορεί να έχει θετικές επιπτώσεις και στις αναπτυσσόμενες χώρες. Χαίρομαι πάρα πολύ που περισσότερες πολιτικές ομάδες το δέχονται αυτό. Ευχαριστούμε πολύ. Ας δώσουμε πάλι το λόγο στην κυρία Ρέντινγκ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα καταλάβατε από τις παρεμβάσεις αυτές ότι ε, υπάρχουν πολλά σημεία σύγκλησης. Υπάρχουν όμως ακόμα κάποια εκκρεμή ζητήματα τα οποία πρέπει να διευθετήσουμε. Και αυτό ακριβώς πρόκειται να κάνουμε στο μέλλον. Και μάλιστα ήδη από την επόμενη συνεδρίαση αύριο θα συναντηθώ με τους σκιώδεις συγητές και θα προσπαθήσουμε να θεραπεύσουμε όλα αυτά τα σημεία απόκληση, τα οποία δεν είναι πολλά. Νομίζω θα καταφέρουμε να καταλήξουμε σε μια πραγματική συμφωνία. Πρέπει λοιπόν να καταφέρουμε να προτείνουμε κάτι βιώσιμο και έγκυρο όσον αφορά τη δική μας Επιτροπή για να καταφέρουμε να ψηφίσουμε τελικά τον Δεκέμβριο. Χαίρομαι πάρα πολύ για τις επικοδομητικές αυτές παρεμβάσεις που άκουσα από τις 9 επιτροπές οι οποίες γνωμοδοτούν, η κάθε μία προφανώς για τον δικό της τομέα αρμοδιότητας. Νομίζω ότι οι γνωμοδοτήσεις αυτές πραγματικά μας βοηθούν και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να τις συμπεριλάβουμε και αυτές στην τελική έκθεση. Πρόκειται για μια σημαντική εργασία που έχουν κάνει οι συνάδελφοί μας στις άλλες επιτροπές. Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζω να ελπίζω πως θα καταφέρουμε ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα. Σας ευχαριστώ πολύ κλείνει με αυτό το σημείο της ημερησίας διάταξης και περνάμε στο σημείο 17. Έχουμε τον Υπουργό Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Λουξεμβούργου, Ζαν Άθελμπορν, ο οποίος ήρθε για να μας ενημερώσει για τις ε, δραστηριότητες της Λουξεμβουργιανής Προεδρίας και τις επιτυχίες της. Ε, καταφέραμε χθε λοιπόν να ολοκληρώσουμε μια πάρα πολύ σημαντική συμφωνία η οποία θα αποτελέσει προηγούμενο και για μελλοντικές ε, συμφωνίες. Ωστόσο, δεν έχει τελειώσει ακόμα η Προεδρία του Λουξεμβούργου. Έχουμε ακόμα τον Αϊρόμπι μπροστά μας και είμαστε ε, όλοι πολύ... Ε, και έχουμε όλοι μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει. και πώς ε, θα δρομολογηθούν οι υπόλοιπε ε, διαπραγματεύσεις. Έχετε το λόγο κυρία Φίλμπον. Λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ Μπέντ. Είναι μεγάλη τιμή για μένα το ότι είμαι μαζί σας για μια ακόμη φορά στην σημαντική επιτροπή σας. Εφόσον μου το επιτρέπετε λοιπόν θα χρειαστώ λίγο χρόνο για να σας παρουσιάσω αναλυτικά το που βρισκόμαστε στον τομέα του διεθνούς εμπορίου. Όταν είχα έρθει εδώ τον μήνα Ιούλιο, θεώρησα ότι η Προεδρία αυτά είναι η πρώτη Προεδρία μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας, αυτό ήταν ένα έκτακτο θέμα, είχε να αντιμετωπίσει άλλα σημαντικότερα θέματα και στον τομέα της εμπορικής πολιτικής οι ερωτήσεις δεν τίθενται με τον ίδιο υπαρξιακό τρόπο που τίθενται σε άλλους τομείς, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η εμπορική πολιτική περιορίζεται στην απλή λογική της προστασίας των επενδύσεων ή των τελωνιακών λασμών κτλ. Ήδη τον Ιούλιο στην πρώτη επαφή έδωσα το παράδειγμα της Τινησίας για τα θετικά αποτελέσματα, για να δώσω το παράδειγμα των θετικών αποτελεσμάτων μιας ε, συμπεριληπτικής εξωτερικής πολιτικής υπεύθυνη μέσω όλων των μορφών εμπορίου. Γι' αυτό χαίρομαι που οι διαπραγματεύσεις με την Τινησία για μια συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών ξεκίνησαν στις 13 Οκτωβρίου και ο πρώτος γύρος των επαφών έγινε αμέσως μετά ήδη. Αυτό δείχνει τον τρόπο στήριξης της Ευρώπης σε μια χώρα που δυσκολεύεται να επανεκκινήσει την οικονομία της, για να προτείνει στον πληθυσμό της καλύτερες και μεγαλύτερες προοπτικές. Οι επανειλημμένες τρομοκρατικές επιθέσεις αποδεικνύουν ότι η Ευρώπη θα πρέπει να είναι αλληλέγγυα με το είναι χώρες της γειτονίας της. Το Συμβούλιο είναι και αυτό διαθέσιμο να μπει σε τριμερή διάλογο μαζί σας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σε σχέση με τις επιπλέον ποσότητες ελαιολάδου που προτείνει να εφαρμόσει ήδη από την 1η Ιανουαρίου του 2016. Τώρα, θα έλεγα ότι συνολικά υπάρχουν αρκετά θέματα στα οποία τα αποτελέσματα είναι καλά. Υπάρχουν κάποιες άλλες ερωτήσεις όπου παρά τις προσπάθειες τις οποίες κάναμε δεν πετύχαμε τους στόχους τους οποίους είχαμε θέσει συνειδητοποιώντας τις απαιτήσεις όλων των εμπλεκομένων στον τομέα της διαφάνειας, εμείς συνεχίζουμε τον τακτικό διάλογο μαζί σας και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως φυσικά και με την κοινωνία των πολιτών. Εκπρόσωποι της Προεδρίας ε, πήραν μέρος σε όλες τις συνεδριάσεις της Επιτροπής ΙΝΤΑ, ε, άκουσαν προσεκτικά τους ευρωβουλευτές, ε, τις ομάδες τους ε, πήραν μέρος σε συζητήσεις με την κοινωνία των πολιτών, της ΜΚΟ και τους εκπροσώπους οικονομικών επιχειρηματικών κύκλων. Έτσι λοιπόν και σε επίπεδο πολυμερές και σε επίπεδο τομεακό, βιομηχανία, ανθρώπινα δικαιώματα κτλ. Προσπαθήσαμε με την Επιτροπή σας Πρόεδρε να κατευθύνουμε τις κοινέ μας ε, ε, ενασχολήσεις τους τελευταίους μήνες. Τώρα για τη νέα ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Εμπόριο της 14ης Οκτωβρίου δεν χρειάζεται να επανέλθω. Τα είχατε συζητήσει με την Επίτροπο Μάλστρομ και μαζί μας το Συμβούλιο. Το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων Εμπορίου υιοθέτησε συμπεράσματα γύρω από αυτό το θέμα που πετύχαμε να καταλήξουμε σε αυτά πολύ γρήγορα. Να αναφερθώ σε ένα θέμα εδώ σύντομα που σας ενδιαφέρει πολύ, δηλαδή τη δημοσίευση της εντολής του Συμβουλίου. Εγώ είμαι υπέρ της διαφάνειας προσωπικά και οσδήποτε θα πρέπει να είναι σε θέση να πάρει μέρος στις οδηγίες για την διαμόρφωση της εντολής. Και από ό,τι κατάλαβα ένα σύστημα πληροφορικό θα επιτρέψει πάρα πολύ σύντομα να υπάρχει ηλεκτρονική επικοινωνία ανάμεσα στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Αυτό ελπίζω ότι θα λύσει τις δυσκολίες που υπάρχουν σήμερα ανάμεσα στα δύο όργανα για το συγκεκριμένο θέμα. Να πω επίσης ότι οι αποφάσεις για την δημοσίευση της συγκεκριμένης κάθε φορά εντολής θα λαμβάνονται κατά περίπτωση είναι ένα θέμα το οποίο θα έλεγα που απαιτεί ομοφωνία στο Συμβούλιο. Πέραν τούτου ε, είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει και το έχουμε ήδη κάνει αποστέλλοντας ε, τις, ε, τα στάδια των διαπραγματεύσεων για τη Διεθνή Σύμβαση για τα, για τα περιβαλλοντικά αγαθά κατά κάποιο τρόπο. Θα υπάρξει συνάντηση της αρμόδιας ομάδας στις 15 ε, με 18 Δεκεμβρίου στο Ναϊρόμπι. Ε, απαιτείται 15 ε, υπουργοί να είναι παρόντες για να μπορέσουν να υπάρξουν αποφάσεις. Θα προσπαθήσουμε να αξιολογήσουμε τη γενικότερη σφαιρική ισορροπία που θα μπορούσαμε να δεχτούμε σε σχέση με την ανάπτυξη, τον ανταγωνισμό και τις υποδομές έτσι λοιπόν στο Ναϊρόμπι θα πρέπει να δούμε τι θα αποφασίσουμε και για την επόμενη περίοδο. Το πακέτο για το Ναϊρόμπι περιλαμβάνει τμήματα του πακέτου Ντόχα για την ανάπτυξη και εκεί τα αποτελέσματα, ή μάλλον οι προοπτικές για να πετύχουμε αποτελέσματα ήταν αρκετά καλά υποσχόμενες σε σχέση με την ανάπτυξη επαναλαμβάνω ιδιαίτερα για τις λιγότερο προχωρημένες χώρες. Η εμπλοκή και δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέρ των χωρών αυτών θα παραμείνει ισχυρή και νομίζω ότι θα έχουμε να παίξουμε ένα καθοριστικό ρόλο. Έχει υπάρξει σημαντική πρόοδο σε δύο από τα τέσσερα θέματα του Μπαλί ε, σε σχέση με τις χώρες προέλευσης, αλλά για το βαμβάκι, για την πρόσβαση στις αγορές και την έλλειψη ε, περιοριστικού ποσοτικού είναι κάτι το οποίο δεν έχει ακόμα λυθεί σχετικά τώρα με την ειδική και διαφοροποιημένη μεταχείριση είναι ένα θέμα που απαιτεί πολύ περισσότερο λεπτομερή συζητήσεις. Ο ανταγωνισμός της εξαγωγής στον γεωργικό τομέα έχει σαν στόχο να υπάρξει μια μεγαλύτερη θα έλεγα πειθαρχία ε, για την ενίσχυση των γεωργών, δηλαδή τις επιδοτήσεις για τις εξαγωγές, ε, τις πιστώσεις εγγύησης, τις ε, εξαγωγικές κρατικές επιχειρήσεις και την διεθνή επισητιστική βοήθεια. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι απαραίτητο τα αποτελέσματα να περιλαμβάνουν τα θέματα τα τέσσερα ε, του ανταγωνισμού για τις εξαγωγές και καταθέσαμε μια κοινή πρόταση με Βραζιλία, Παραγουάη, ε, Νέα Ζηλανδία, Περού και Ουρουγουάη στις 16 Νοεμβρίου του 2015. Υπάρχει πιθανότητα θετικών αποτελεσμάτων σε σχέση και με τους κανόνες αντιεπιδοτήσεων, αντι-dumping, περιφερειακών συμφωνιών, αλλιευτικών συμφωνιών και διακανονισμός παροχής υπηρεσιών. Σχετικά τώρα με τους τρεις, την ομάδα των τριών πρέσβεων, ο διευθυντής του ΠΟΕΟ κ. Ασεβέντο παρουσίασε πριν λίγο καιρό μια πρόταση συμβιβαστική για τα διαδικαστικά που συνεχίζουν να είναι υποσυζήτηση στη Γενέβη. Ε, μέχρι την τελευταία στιγμή θα γίνονται διαπραγματεύσεις και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της έτσι ώστε ο ΠΟΕ να βγει ενισχυμένο από αυτή την υπουργική διάσκεψη η οποία κατ' εμέ θα πρέπει να επιτρέψει να γίνει μια σοβαρή συζήτηση και για τη συμπερίληψη νέων θεμάτων στις πολυμερείς συζητήσεις ε, διατηρώντας βέβαια τον κεντρικό χαρακτήρα θεμάτων όπως η ανάπτυξη γενικότερα, η ζάχαρη, το καθεστώς της ζάχαρης κτλ. Αφού μελέτησα το ψήφισμά σας της προηγούμενης πέμπτης μπορώ να πω ότι έχουμε κοινού στόχους ε, για το ζήτημα αυτό. Συνάντησα τους γενικούς διευθυντές του ΠΟΕ στην ε, Κωνσταντινούπολη στα πλαίσια επίσης της συνόδου του G20 που έλαβε χώρα στην Τουρκία και παρουσία της Εσίλια Μάλστρομ τους έδωσα την ε, εντολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, όσον αφορά την διευκόλυνση των ε, διαπραγματεύσεων για το ζήτημα της σύναψης συμφωνιών ελεύθερου εμπορίου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω γι' αυτό τη δική σας Επιτροπή και γενικότερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που βοήθησε την σύντομη έγκριση της συμφωνίας αυτής. Όσον αφορά τώρα το Συμβούλιο, τους τελευταίους μήνες ασχοληθήκαμε περισσότερο με, τις, ε, με τους αποκλεισμούς όσον αφορά τις ε, υπηρεσίες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ουσιαστικά λάβαμε υπόψη μας όλες τις ανάγκες των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών. Επίσης ασχοληθήκαμε με τον αποκλεισμό των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών πρόσφατα και στα τέλη Ιουλίου στην ε, αρμόδια επιτροπή του ΠΟΕ καταβλήθηκαν όλες οι απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ζήτημα αυτό. Στην Υπουργική Διάσκεψη του Ναϊρόμπι ήμασταν σε θέση να πούμε ακριβώς ποιες ήταν οι προτιμήσεις που μπορούσαν να προωθήσουν οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωση στον τομέα των υπηρεσιών για τις λιγότερες αναπτυγμένες χώρες. Στα πλαίσια της 10ης Υπουργικής Διάσκεψης του ΠΟΕ στο Ναϊρόμπι, ελπίζουμε και σε πολιτικό επίπεδο να πετύχουμε μια πολυμερή συμφωνία όσον αφορά τα περιβαλλοντικά αγαθά. Η συμφωνία αυτή εγγράφεται με τη σειρά της σε μια μεγαλύτερη συνεκτικότητα της εμπορική μας περιβαλλοντικής, βιομηχανικής πολιτικής και πολιτικής καινοτομίας. Η συμφωνία αυτή θα είναι πάρα πολύ σημαντική στα πλαίσια των κλιματικών διαπραγματεύσεων της COP21 στο Παρίσι, καθώς επίσης και στα πλαίσια της προηγικής διάσκεψης του ΠΟΕ στο Ναερόμπι. Στη συμφωνία αυτή μπορούν να συμμετέχουν όλα τα κράτη-μέλη του ΠΟΕ που θέλουν να συνταχθούν με τη φιλόδοξη αυτή προσπάθεια που θα έχει σημαντικές βιομηχανικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές επιπτώσεις, καθώς επίσης και μια τεράστια συμβολική σημασία για την Ευρώπη και τους εταίρους της. Όσον αφορά τώρα άλλες ε, πολυμερείς ε, διαπραγματεύσεις θα ήθελα να αφαιρθώ στην ολοκλήρωση της ε, συμφωνίας όσον αφορά την ε, τεχνολογία της πληροφορικής. ITA. Αυτή θα ολοκληρωθεί πιστεύω μέχρι την υπουργική διάσκεψη του Ναϊρόμπι. Όσον αφορά τώρα τι διαπραγματεύσει για τη συμφωνία TISA, την οποία καλύψατε, αν δεν κάνω λάθο, πριν από λίγο, η Προεδρία του Λουξεμβούργου παρακολούθησε εκ του σύνεγγυ τι διαπραγματεύσει στα πλαίσια του Συμβουλίου. Είναι πολύ σημαντικό η συμφωνία αυτή να καταφέρει να οδηγήσει οικονομική τόνωση και αύξηση της απασχόλησης. Θα πρέπει όμως να βασίζεται σε κανόνες οι οποίοι δεν θα οδηγούν σε καμία διακριτική μεταχείριση. Και Γι' αυτό το λόγο η Προεδρία του Λουξεμβούργου θέλει να διασφαλίσει ότι είναι πολύ σημαντικό τα κράτη-μέλη να εξακολουθούν να μπορούν να νομοθετούν. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο είναι πολύ σημαντικό να αποκλείονται από τη συμφωνία αυτή οι δημόσιες υπηρεσίες, οι υπηρεσίες κοινή ωφελίας. Υποστηρίξαμε με επικοδοματικό τρόπο όλου τους συμμετέχοντες στι συζητήσει αυτέ, αυτές, με συγχωρείτε, και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προκειμένου να έχουμε νέους κανόνες για τις υπηρεσίες, οι οποίοι όμως θα σέβονται το κοινοτικό και και θα δίνουν νέες δυνατότητες στους παρόχους υπηρεσιών. Απότερος στόχος είναι να καταλήξουμε σε όσο το δυνατόν περισσότερες χώρες οι οποίες να συμμετέχουν σε αυτή τη συμφωνία. Μόνο κατά αυτόν τον τρόπο αυτή η συμφωνία μπορεί να γίνει πραγματική πολυμερής πλειονοτική συμφωνία. Είναι πολύ σημαντικό επίσης ε, να τονίσουμε τις πολύ σημαντικές προσπάθειες που έκανε η δική σας επιτροπή και η Vivian Redding που προέρχεται και αυτή από το Λουξεμβούργο. Συνεχίσαμε επίσης στα πλαίσια του Συμβουλίου όλες τις προσπάθειες προκειμένου να προσχωρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τη διαφάνεια όσον αφορά την ε, διαιτησία ανάμεσα στα κράτη και τις επιχειρήσεις. Γνωρίζετε ότι υπάρχει πρόβλημα προς αυτό. Εμείς θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να καταδείξει ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει ένα ανώτατο επίπεδο διαφάνειας και θα πρέπει να εφαρμοστούν το συντομότερο δυνατό οι προβλεπόμενοι κανόνες από το CDIE στα πλαίσια των διαδικασιών διαιτησίας για τα δύο ένδικα μέρη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν από τους σημαντικότερους παράγοντες ε, στην ε, σύναψη της συμφωνίας αυτής και είναι πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να διασφαλίσουμε στα πλαίσια αυτής της συμφωνίας την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άλλωστε μιλάμε για μια πολυμερή συμφωνία στην οποία συμμετείχε εξ αρχής η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, τελευταίους μήνες προσπαθήσαμε με τρόπο ραλιστικό και επικοδομητικό σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βρούμε πρακτικές λύσεις προκειμένου να βγούμε από το υφιστάμενο διέξοδο που έχουμε, μολονότι έχει σημειωθεί πρόοδος. Για πάρα πολλά σημεία δεν υπάρχει ακόμα κοινή συμφωνία όλων των κρατών μελών στο Συμβούλιο και δυστυχώς δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμα να προσχωρήσει σε αυτή τη σύμβαση. Αυτό πραγματικά είναι λυπηρό και ουσιαστικά έχει αρνητικές επιπτώσεις στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα συνεχίσουμε να καταβάλουμε λοιπόν προσπάθειες προκειμένου να καταλήξουμε σε μία λύση, να συμφωνήσουμε όλα τα κράτη-μέλη και να καταφέρουμε να προσχωρήσουμε τελικά σε αυτή τη συμφωνία των Ηνωμένων Εθνών για τη διαφάνεια. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να αφαιρθώ τώρα στις διμερείς εμπορικές διαπραγματεύσεις που διεξάγει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τρίτες χώρες. Κατά τη διάρκεια της δικής μας της Προεδρίας προσπαθήσαμε να καταλήξουμε σε μία συμφωνία, μια, σε μία πρόοδο, αν θέλετε, στις διαπραγματεύσεις που γίνονται για το TTIP. Τους τελευταίους, οι τελευταίοι μήνες ήταν ιδιαίτερα καθοριστικοί, καθότι προσπαθήσαμε να καθορίσουμε ποιο δρόμο θα πρέπει να ακολουθήσουμε για τα πιο πολιτικά, θέλετε, ζητήματα. Το ζήτημα των, τα αριθμιστικά ζητήματα, ο εξεχρονισμός του συστήματος προστασίας των επενδύσεων, καθώς επίσης και οι δημόσιες συμβάσεις. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο. Αυτή τη φορά βάλαινε και στο, στην πλευρά των Αμερικάνων. Ξέρω ότι ο μηχανισμό ISDS και η μεταρρύθμισή του μα απασχόλησε ιδιαίτερα του τελευταίου μήνε, επίλυση διαφορών επενδυτή κράτου. Στην αρχή του έτου, εσεί, κύριε Πρόεδρε, με ορισμένου υπουργού εμπορίου τη Γερμανία, τη Γαλλία, τη Σουηδία, τη Δανία, των κάτω χωρών και του Λουξεμβούργου, προσπαθήσαμε από κοινού να ασχοληθούμε με το ζήτημα αυτό για να προτείνουμε μια μεταρρύθμιση του συστήματος αυτού. Το Συμβούλιο όμω και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μελέτησαν και αυτά το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το TTIP, το οποίο εγκρίνατε εσείς τον Ιούλιο. Λαμβάνουμε λοιπόν υπόψη μας τις συστάσεις που κάνετε και το περιεχόμενο του ψηφίσματος αυτού. Το Σεπτέμβριο τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε μια πρόταση όσον αφορά ένα νέο σύστημα διευθέτηση των διαφορών μεταξύ επενδυτών και κράτου, ένα investment court system όπω ονομάζεται ECS. στόχος της νέας αυτής πρόταση είναι να έχουμε ένα ανώτερο επίπεδο διαφάνειας και να μπορούμε να διασφαλίσουμε τις αρμοδιότητες και τα δικαιώματα των κρατών μελών να μπορούν να εξακολουθούν να νομοθετούν και να οριοθετούν τον τρόπο με τον οποίο θα αναλαμβάνουν δράση οι επιχειρήσεις, κυρίως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το νέο αυτό σύστημα προβλέπει τη δημιουργία ενός αμερόληπτου διαφανούς συστήματος το οποίο θα απασχολεί δικαστές οι οποίοι θα διορίζονται δημόσια και θα προβλέπει μάλιστα και ένα σύστημα υποβολής θέσεων. Θα υπάρχει και ένα εφετείο. Καταλαβαίνετε λοιπόν το νέο αυτό σύστημα διαφέρει πάρα πολύ από το υφιστάμενο σύστημα ISDS. Είναι σημαντικό όμως να καταφέρουμε να προστατεύσουμε και τους Ευρωπαίους επενδυτές και να μπορούμε να διευθετούμε με τον πιο αντικειμενικό τρόπο τις διαφορές που θα προκύψουν. Η Λουξεμβουργιανή λοιπόν Προεδρία προσπάθησε να πετύχει μια συμφωνία στα πλαίσια της αρμόδιας επιτροπής προκειμένου να επιτρέψουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσημα να συζητήσει το ζήτημα αυτό με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το σχετικό έγγραφο κοινοποιήθηκε στις αρχές Νοεμβρίου στις Αμερικανικές Αρχές. Το νέο αυτό σύστημα θα μπορούσε να αποτελέσει μάλιστα παγκόσμιο σημείο αναφορά όσον αφορά την προστασία των επενδύσεων. Στο Συμβούλιο της προηγούμενης Παρασκευής είπαμε ότι εκτιμούμε θετικά την προσέγγιση αυτή που υιοθετεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καταβάλουμε λοιπόν προσπάθειες προκειμένου όντως να υπάρχει πρόσβαση σε κάποια εμπιστευτικά κείμενα στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων TTIP. Το ζήτημα αυτό θα διευθετηθεί πολύ σύντομα. Ο Μάικ Φρούμαν έδωσε επί της αρχής ε, τη δική του σύμφωνη γνώμη προκειμένου να δημιουργηθεί μια αίθουσα ανάγνωσης όπου θα μπορούσε κανείς να διαβουλεύεται τα εμπιστευτικά αυτά έγγραφα. Και αυτό αποτελεί πολύ σημαντικό επίτευγμα όσον αφορά το ζήτημα της διαφάνειας και αυτό έχει αποτελέσει προτεραιότητα τόσο για σας όσο και για μας. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να τονίσω και την εξαιρετική εργασία που έγινε από την Επίτροπο κυρία Βάλστρομ, η οποία δείχνοντας ανοιχτό πνεύμα, διαλλακτικότητα και επικοδομητική στάση, κατέβαλε συνεχείς προσπάθειες προκειμένου να αυξηθεί το επίπεδο διαφάνειας διαπραγματεύσεων του TTIP. Επίσης, το ίδιο ανοιχτό πνεύμα συνεχίζεται και ο διάλογος με όλους εμπλεκόμενους φορείς και η Προεδρία του Λουξεμβούργου οργάνωσε μία συνεδρίαση στις Βρυξέλλες πρόσφατα για το TTIP, όπου για πρώτη φορά είχαμε και κοινωνικούς εταίρους από τα 28 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χαίρομαι πάρα πολύ που από ό,τι φαίνεται είναι πλέον δυνατό να συζητούμε για το TTIP με έναν τρόπο πιο ισότιμο και ανοιχτό. Όσον αφορά τώρα τις εξελίξεις από την Αμερικανική πλευρά, το ESTR στις 5 Νοεμβρίου δημοσιοποίησε την τελική σχεδόν εκδοχή της συμφωνίας για τον ειρηνικό, ο πρόεδρος Ομπάμα είπε επίσης ότι θέλει να προωθήσει την σύναψη συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρετε όμως ότι το Κογκρέσο έχει στη διάθεσή του 90 μέρες για να εξετάσει το έγγραφο προτού το εγκρίνει επισήμως. Αυτό προβλέπεται στα πλαίσια της νομοθεσίας Fast Track που ενέκρινε το Κογκρέσο νωρίτερα φέτος. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την εξέταση του κειμένου αυτού από το Κογκρέσο. Δεν πρόκειται πριν από τον Απρίλιο το Μάιο του 2016 να υπάρξει ψηφοφορία στο Αμερικανικό Κογκρέσο. Και όλα αυτά επηρεάζονται επίση και από την προεκλογική καμπάνια στι ΗΠΑ. Σε κάθε περίπτωση πάντω θέλουμε να, καλύξουμε, να καταλήξουμε σε μια φιλόδοξη συμφωνία μέχρι τα τέλη του επόμενου έτου αλλά καταλαβαίνετε ότι επηρεαζόμαστε πάρα πολύ και από το υφιστάμενο χρονοδιάγραμμα αυτή τη στιγμή. Όπω είπα και στην πρώτη μου παρέμβαση στη δική σα την Επιτροπή, θέλουμε αυτή τη στιγμή να ανταποκριθούμε σε αυτόν τον πολυμερή κόσμο, ο οποίο αρχίζει και διαφαίνεται όλο και περισσότερο, οπότε είναι πολύ σημαντικό να έχουμε μια ποιοτική συμφωνία με τι Ηνωμένε Πολιτείε. Η συμφωνία αυτή θα οδηγήσει σε μια καλύτερη κατανόηση των της υφιστάμενης κατάστασης όσον αφορά το εμπόριο και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Πολλές φορές μας δίνει την εντύπωση ότι δεν έχουμε τον απόλυτο έλεγχο όσον αφορά τη συμφωνία ΣΕΤΑ. Εδώ δεν έχω να πω σπουδαία πράγματα. Ο νομικός έλεγχος Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι σε εξέλιξη. Είμαι όμως πεπισμένος ότι θα πρέπει το συντομότερο δυνατό και αν δεν κάνω λάθος αυτό ήδη έχει ξεκινήσει, η Σεσίλια ήδη είναι σε επαφή με τη νέα Υπουργό, του Καναδά. Να συζητήσουμε λοιπόν το συντομότερο δυνατό την ε, συμφωνία αυτή και ιδίω όσον αφορά το κεφάλαιο εκείνο που έχει να κάνει με την επίλυση των διαφορών επενδυτή κράτου. Μια άλλη προτεραιότητα τη Λουξεμβριανή Προεδρία είναι οι ε, διμερεί συμφωνίε. Εντείναμε τι συζητήσει για να έχουμε μια φιλόδοξη συμφωνία εμπορικών συναλλαγών με την Ιαπωνία. Οι ε, συζητήσει που έλαβαν χώρα φέτος δεν κατέληξαν στο ευκαιρό αποτέλεσμα, μάλλον ότι ο Υπουργό Σαμπέ και ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ άσκησαν ιδιαίτερη πίεση. Ήδη την προηγούμενη Παρασκευή συζητήσαμε το ζήτημα αυτό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε ένα νέο χρονοδιάγραμμα για να καταλήξουμε τελικά σε συμφωνία το 2016. Στην ίδια περιοχή του κόσμου χαίρομαι πάρα πολύ που η Ευρωπαϊκή Ένωση ολοκλήρωσε μια διαδικασία επικύρωση συμφωνίας εμπορικών συναλλαγών με την Κορέα μετά από πέντε ολόκληρα χρόνια. Έχετε δίκιο κύριε Πρόεδρε. Ναι, αλλά πάνω από πέντε χρόνια κράτησαν οι ανάλογε διαπραγματεύσει μεταξύ Ασίας και Ηνωμένων Πολιτειών. Ήδη από τα μέσα Δεκεμβρίου ισχύει λοιπόν αυτή η νέα συμφωνία προβλέπεται η δυνατότητα εξυγχρονισμού της συμφωνίας αυτής με την κορεατική πλευρά στα πλαίσια του Συμβουλίου. Επίσης, κατά τη διάρκεια της δικής μας της Προεδρίας, καταφέραμε να ολοκληρώσουμε τις διαπραγματεύσεις ε, για μια εμπορική συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, και του Βιετνάμ. Η συμφωνία αυτή έχει να κάνει με την απελευθέρωση των δασμών, το άνοιγμα των αγορών, την τήρηση όλων των υποχρεώσεων όσον αφορά τις, τα πνευματικά δικαιώματα. Χαίρομαι πάρα πολύ που το Βιετνάμ, το οποίο εδώ και πάρα πολλά χρόνια αποτελούσε ε, χώρα στόχο για τα επίσημα προγράμματα αναπτυξιακής βοήθειας κατάφερε τελικά να φτάσει στο σημείο να συνάψει μια τόσο φιλόδοξη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών. Επεξεργαζόμαστε το τμήμα των επενδύσεων. Η βιετναμική πλευρά και ο κύριος Γιούνκερ ήδη αυτή την εβδομάδα θα καταφέρουν να ολοκληρώσουν το σχετικό αυτό κεφάλαιο. Ε, Γενικότερα λοιπόν και μιας και το διαπιστώσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα οι προσπάθειες εμβάθυνσης των οικονομικών σχέσεών μας με τα μέλη του ΑΣΕΑΝ και σε επίπεδο διπεριφερειακό και σε επίπεδο κατά περίπτωση ε, διμερές ε, έχουν αρχίσει να καρποφορούν. Ξεκινήσαμε διαπραγματεύσεις με τις Πιλιππίνες και ελπίζω ότι και θα προβλεφτούν διαπραγματεύσεις το 2016 με την Ινδονησία. Είμαστε έτοιμοι για να ξεκινήσουμε και στις συζητήσεις για τη Μαλαισία και την Ταϊλάνδη γνωρίζοντας ότι είναι δύσκολο για τη Μαλαισία και αδύνατο προς το παρόν για την Ταϊλάνδη. Η συμφωνία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Κίνα για μια αναπτυξιακή συμφωνία συνεχίστηκαν κατά τη διάρκεια του 2015. Είναι προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επανεξισορρόπηση αμοιβαίως ωφέλιμη των σχέσεων με την Κίνα. Το Συμβούλιο συνεχίζει να παρακολουθεί από κοντά τις προσπάθειες της Επιτροπής και υπογράμμισε την μεγάλη σημασία που έχει για τους διαπραγματευτές να εντατικοποιήσουν τις προσπάθειές τους για να καταλήξουν με την κινέζικη πλευρά στον καθορισμό της ευέλειας της συμφωνίας και να καταλήξουν σε ένα κοινό κείμενο σαν βάση για τις περαιτέρω διαπραγματεύσεις. Στα πλαίσια αυτά συζητήσαμε και την επενδυτική συμφωνία με τη Μιανμάρ για να δώσουμε στην επιχειρηματικότητά μας περισσότερες δυνατότητες ασφάλειας, εγγύησης των επενδύσεων και μείωσης των εμποδίων σε αυτή τη χώρα υπομετάβαση, μια μετάβαση την οποία θα πρέπει να στηρίξει η Ένωση όπως μπορεί. Εάν για τις συμφωνίες αυτές ε, είναι κεντρικό σημείο το θέμα των επενδύσεων και της εγγύησης των επενδύσεων, θα συνεχίσουμε να είμαστε πολύ φιλόδοξοι και στον τομέα των μεταφορών και στον τομέα της αηφορίας Πρέπει εδώ να αναφέρουμε και τις συμφωνίες με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Ελπίζουμε να ξεκινήσουμε σύντομα εμπορικές διαπραγματεύσεις. Το Συμβούλιο έχει δώσει την έγκρισή του για το λεγόμενο σκούπινγκ μέχρι το τέλος του επόμενου χρόνου ε, για τη, για τη συμφωνία με αυτές τις δύο χώρες. Δεν αναφέρθηκε στο Μερκοσούρ. Εκεί παρά τις προσπάθειές μας δεν έχουν καταλήξει οι διαδικασίες οι συζητήσεις οι οποίες έγιναν μέχρι την προηγούμενη Τετάρτη ε, οδήγησαν σε συζητήσεις πάρα πολύ ειλικρινείς και άμεσες. Και όταν λέω άμεσες καταλαβαίνετε τι έγινε. Το λέω διπλωματικά. Αυτό επέτρεψε στην Επίτροπο Μάλστρομ να καταλάβει τι πιστεύουν οι διάφορες αντιπροσωπείες οι εθνικές. Πάντως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει τις προσπάθειες λαμβάνοντας υπόψη τα αμυντικά αλλά και επιθετικά της συμφέροντα αυτό θα πρέπει να γίνει όμως με ισχυρά θεμέλια. Τώρα για το ειδικό θέμα της μειωμένης κάλυψης των ε, δασμολογικών γραμμών, εκεί υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στις εθνικές συνιστώσεις. Τώρα για τη γειτονία. Ε, θα έλεγα ότι η κρίση των προσφύγων απέδειξε ότι οι διάφορες πολιτικές πρωτοβουλίες στις γειτονικές μας χώρες θα πρέπει να είναι σφαιρικές και συνεκτικές. Γι' αυτό και χαιρετίζω τη συμφωνία στην οποία καταλήξαμε και ανέφερε ο Πρόεδρος χθε στον τριμερή διάλογο για τα Δυτικά Βαλκάνια, τα αυτόνομα μέτρα. Ε, χαίρομαι που καταλήξαμε σε μια πραγματιστική θέση που θα, επι... θα, θα δώσει τη δυνατότητα επιβίωσης της οικονομίας αυτών των περιοχών. Νομίζω ότι και η συμφωνία με την Ουκρανία θα τεθεί σε λειτουργία την 1η Ιανουαρίου του 2016 σε αυτό το πλαίσιο εμπειρογνώμονες από την Ένωση, την Ουκρανία και τη Ρωσία συνεχίζουν ακόμα και σήμερα τις τριμερείς επαφές τους. Δεν θα πρέπει να έχουμε πάρα πολλές ελπίδες βέβαια, έτσι ώστε η συμφωνία αυτή να μην οδηγήσει σε μια χειροτέρευση της οικονομικής και πολιτικής κατάστασης. Ο διάλογος θα πρέπει να συνεχιστεί σεβόμενοι τα συμφέροντα της κάθε χώρας και περιοχής και η κυρία Μάστρομ είπε ήδη ότι ακόμα και αν το πρόβλημα δεν λυθεί μέχρι την 1η Ιανουαρίου η εμπλοκή μας ε, στον διάλογο με τη Ρωσία θα συνεχιστεί. Όπως είχα εξηγήσει και την τελευταία φορά που ήρθα εδώ θα συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε τις κατά προτίμηση εμπορικές μας σχέσεις με τους αφρικανικούς εταίρους. Οι συμφωνίες εταιρικών σχέσεων ενισχύουν τις σχέσεις μας σε νέα βάση με την Αφρικανική Ήπειρο. Μια Ήπειρο η οποία έχει να αντιμετωπίσει πάρα πολλές δυσκολίες αλλά έχει και πάρα πολλές ευκαιρίες. Το εμπόριο δεν θα πρέπει να χρησιμεύσει μόνο στην οικονομική ανάπτυξη των εταίρων μας αλλά και σε μια αμοιβαία κατανόηση και στην κοινωνική και περιβαλλοντική πρόοδο στα πλαίσια μιας συνεχούς και ισχυρής εταιρικής σχέσης. Νομίζω ότι αυτό αποδεικνύεται από τις επιμέρους πολιτικές μας. Η υπογραφή της συμφωνίας με την κοινότητα του νοτίου τμήματος της Αφρικής, της Μεσημβρινή Αφρική δηλαδή, θα ολοκληρωθεί τον Απρίλιο του 2016 και αυτό θα οδηγήσει στην ενίσχυση των οικονομικών σχέσεων με όλες τις χώρες αυτές στο νότιο τμήμα της Αφρικής. Πριν περάσω στο νομοθετικό κομμάτι, να αναφερθώ και σε κάτι άλλο το οποίο απασχολεί τις χώρες μας στον τομέα της ε, χαλιβουργίας. Η χαλιβουργία στην Ευρώπη αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις και συγκυριακές και διαφορετικές. Καταρχάς υπάρχει υπερπαραγωγή διεθνής, μείωση της ζήτησης και ε, στρεβλές εμπορικές πρακτικές τρίτων χωρών. Υπάρχουν επίσης και εθνικές ενεργειακές πολιτικές που οδηγούν σε υψηλότατο κόστος ενέργειας. Η παραγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντιπροσωπεύει 360.000 άμεσης απασχόλησης. Ε, με πρωτοβουλία της Προεδρίας το θέμα τέθηκε στο Συμβούλιο ήδη και την προηγούμενη Παρασκευή για να βρεθούν μέτρα για να διορθωθεί η κατάσταση αυτή, λαμβάνοντας υπόψη τα μέσα τα οποία μας δίδει η εμπορική πολιτική. Το θύμισα το θέμα αυτό γιατί ο Χάλιβας και για τη δική μου χώρα είναι πολύ σημαντικό θέμα. Και ο Χάλιβας μέσω της ΕΚΑ φυσικά σας θυμίζω ότι μας έφτιαξε όλους εμάς. Και φυσικά από εκεί και πέρα οικοδομήσαμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τελειώνοντας θα ήθελα να αναφερθώ στις διαδικασίες που τρέχουν στον τομέα των συνομοθετικών. Μία πρόταση της ε, Προεδρίας του Λουξεμβούργου είναι η πρόταση κανονισμού για τα ορυκτά προϊόντα από περιοχές συγκρούσεων. Θέλουμε να σπάσουμε το σύνδεσμο ανάμεσα στην εξαγωγή των προϊόντων, στην εξόριξη αυτών των πρώτων υλών ε, και στις επιτόπους συγκρούσεις στις διάφορες χώρες και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πήρε μία απόφαση και τον μήνα Μάιο. Η Λουξεμβουργιανή Προεδρία οδήγησε τις συζητήσεις στο Συμβούλιο, έχουμε προοδεύσει, νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά σε μια τελική θέση και θα μπορέσουμε σύντομα να ξεκινήσουμε τον τριμερή διάλογο. Είμαι ευεπισμένο ότι με τη δική σας υποστήριξη κύριε Πρόεδρε και με το πακέτο το οποίο θα αποστείλουμε και θα μεταφέρουμε μάλλον στους Ολλανδούς διαδόχους μας υπάρχει δυνατότητα έβρεσης λύσης. Δεύτερον, τροπολόγηση του κανονισμού κατά των βασανιστήριων θα υιοθετηθεί από το αυριανό Κορεπέρ της 2 Δεκεμβρίου και ο πρώτος τριμερής διάλογος θα γίνει την επόμενη εβδομάδα στις 10 Δεκεμβρίου. Η Λουξεμβουργιανή Προεδρία πέτυχε το στόχο της έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η εντολή στις διαπραγματεύσεις του Συμβουλίου και η αρχή του τριμερούς διαλόγου. Λυπάμαι που δεν ξεκίνησε ήδη ο τρίλογος ή ο τριμερής διάλογος καλύτερα. Ελπίζω όμως ε, να συνεχιστεί με βάση τις δικές μας προσπάθειες ε, και τις προσπάθειες των Ιταλών και των Λετωνών παλαιότερα. Περιμένετε την απόφαση του Συμβουλίου, την αντίδραση του Συμβουλίου για το Διεθνής ε, για τα λεγόμενα IPR. Στα πλαίσια της συνάντησης της ομάδας του Συμβουλίου <clears throat> το Συμβούλιο κάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει μια νέα πρόταση. Ελπίζουμε λοιπόν από την επόμενη Προεδρία να συνεργαστεί μαζί μας. Κατά τη διάρκεια του γεύματος εργασίας του Συμβουλίου Εμπορίου την προηγούμενη εβδομάδα συζητήσαμε ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα το να δοθεί δηλαδή η ιδιότητα της οικονομίας ε, της αγοράς στην ε, λαϊκή Κίνα. Οι συζητήσει που έγιναν αποδεικνύουν την περιπλοκότητα του θέματος αυτού. Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφασίσει να μην δοθεί αυτόματα η ιδιότητα αυτή, ο χαρακτηρισμός αυτός τον Δεκέμβριο του 2016, τότε η Κίνα θα μπορεί να κάνει έφεση εις βάρος της απόφασης του ΠΟΕ κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια του μηχανισμού ρύθμισης διαφορών. Αντίθετα με άλλους εταίρους που έχουν μια κάποια δυνατότητα ευελιξία σε σχέση με το θέμα αυτό όπως οι Ηνωμένε Πολιτείε και η Ιαπωνία, σε μας απαιτείται για να αλλάξουμε άποψη μια νομική ρύθμιση στα πλαίσια της τακτικής, της κανονικής νομοθετικής διαδικασίας. Συνεπώς έχουμε πρόβλημα χρόνου για να υπάρξει εδώ μια τροπολόγηση σε σχέση με το αντι-dumping. Ξέρετε ότι απαιτούνται 8 με 12 μήνες κατελάχιστον για τη διαδικασία. Λυπόμεθα που το θέμα αυτό ξεκίνησε να συζητείτε πολύ αργά και ελπίζουμε σαν Συμβούλιο να μπορέσουμε μαζί σας να βρούμε μια βιώσιμη λύση σε αυτό το ακαθόδες θέμα το 2016. Η συζήτηση αυτή θα μπορούσε να επηρεάσει και τις θέσεις των κρατών μελών πάνω στο θέμα του εξυγχρονισμού των μέτρων εμπορικής άμυνας. Όπως ξέρετε τα κράτη-μέλη διαφωνούν σε σχέση με τις νομικές ρυθμίσεις και το Λουξεμβούργο θα συνεχίσει την προσπάθεια για μια ενδιάμεση συνενετική λύση η Προεδρία του Συμβουλίου έκανε πολλή δουλειά έμπας περιπτώσει τους τελευταίους 5-6 μήνες, 5 μήνες γιατί ήταν και ο Αύγουστος στη μέση. Πάντως μπορέσαμε κάποια θέματα να τα φέρουμε εις πέρας και ελπίζω να πετύχαμε τις βασικές μας προτεραιότητες. Είμαι πεπισμένος ότι οι Ολλανδοί συνάδελφοι που θα μας διαδεχθούν θα κάνουν ό,τι μπορούν για να διασφαλίσουν τη συνέχιση της διαδικασίας και για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας στον τομέα των εμπορικών σχέσεων. Σας ευχαριστώ. Λυπάμαι τον Φιντέλ Κάστρο που μιλάει τρεις-τέσσερις ώρες συνέχεια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρία Χαλμπορν, ευχαριστούμε Ζαν. Μας έδωσες μια περιεκτικότατη συνολική εικόνα της, ε, των δραστηριοτήτων της ε, Προεδρίας του Λουξεμβούργου. Τώρα θα δώσω το λόγο στους ευρωβουλευτές έτσι ώστε να κάνουν τις ερωτήσεις του και φυσικά μπορούν να διαβάσουν και όλες τις λεπτομέρειες τα έγγραφα που ε, έδωσες. Ε, βρισκόμαστε υπό πίεση χρόνου, δυστυχώς λοιπόν πρέπει να περιοριστείτε στο ένα λεπτό ο καθένας. Αν θέλετε να πάρετε και απάντηση. Ντάνιελ, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ. Δείξτε παρακαλώ κατανόηση εάν δεν τηρήσω το όριο του ενός λεπτού, διότι ανήκωστε είναι μεγαλύτερη ομάδα εδώ στο Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ καταρχάς πάρα πολύ για την ε, ομιλία σας. Να σας πω ότι το ΕΛΚΑ επιθυμεί να δρομολογηθεί η συμφωνία με την Ουκρανία. Ε, επίσης, ε, θα ήταν καλό... Είναι καλά όλα αυτά που μας είπατε για την ετινησία, όμως θα ήθελα να σταθώ στο ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ζητήσει παράλληλα με την Κίνα να συζητηθεί και με την Ταϊβάν το θέμα της προστασίας των επενδύσεων. Θα θέλετε λοιπόν να μου δώσετε μερικές πληροφορίες παραπάνω για το, ε, για το αν υπάρχει προθυμία να γίνει αυτό στο Συμβούλιο. Έπειτα, Κολομβία και Περού. Αυτή τη στιγμή, αν ε, είμαι καλά πληροφορημένος, η συμφωνία έχει κυρωθεί από 15 κοινοβούλια. Λείπουν όμως ε, κάποια κράτη-μέλη. Τι συμβαίνει εδώ στο Συμβούλιο. Πώς εξελίσσεται η κατάσταση. Θεωρώ επίσης πολύ ενδιαφέρον ε, το ότι το Συμβούλιο στην Συμφωνία ΣΥΤΑ έχει μείνει αρκετά πίσω. Η Συμφωνία ΣΥΤΑ είναι μια πάρα πολύ καλή συμφωνία, όμως αρκετά κράτη-μέλη ζητούν ακόμα περισσότερες βελτιώσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και έτσι παρατείνεται λοιπόν η κυρώση της συμφωνίας. Έπειτα, σχετικά με την νομοθεσία, νομίζω πως ολοκληρώθηκε μόνο ε, ένα νομοθέτημα στην δική σας ε, Προεδρία. Γι' αυτό λοιπόν να διαρωτώ με πώς επιτέλους θα καταφέρουμε να σταματήσουμε όλες αυτές τις καθυστερήσεις στο νομοθετικό έργο στο Συμβούλιο. Στο Κοινοβούλιο υπάρχουν σαφείς κανόνες για τη δεύτερη ανάγνωση τουλάχιστον. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να μου πείτε αν υπάρχουν κάποιοι κανόνες σχετικά με τις αποφάσεις του Συμβούλιο σε πρώτη και δεύτερη ανάγνωση. Ευχαριστώ πολύ. Θα σας απαντήσω πάρα πολύ σύντομα λοιπόν. Ε, Ουκρανία. Ε, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Ε, τώρα, Κίνα και Ταϊβάν. Δεν είμαι εμπειρογνώμων για τις ε, σχέσεις Κίνας και Ταϊβάν, αλλά από ό,τι ξέρω η προτεραιότητα έχει δοθεί στην Κίνα και μετά στην Ταϊβάν. Είναι η λογική ακολουθία των πραγμάτων στο Συμβούλιο. Είναι μια άποψη την οποία δεν συμμερίζομαι κατά ανάγκη, όμως έτσι έχουν τα πράγματα. Τώρα, έχετε δίκιο. Εμείς ως Προεδρία πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τη συμφωνία με το Περού και την ε, Κολομβία, με εκείνα τα κοινοβούλια τα οποία δεν έχουν ε, ακόμα τη συμφωνία και θα μπορούσαμε να ασκήσουμε πίεση στα ε, κράτη. Όμως ε, το παίρνουμε πολύ σοβαρά στο Συμβούλιο αυτό. Τώρα, συμφωνία ΣΥΤΑ. Πιστεύω πως δεν είναι κατά ανάγκη λάθος το σύστημα που ακολουθούμε. Ακόμα και μετά την ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο, Εμεί προσπαθούμε το σύστημα επίλυση διαφορών ε, επενδυτή και κράτους να βελτιωθεί. Κάνουμε ό,τι μπορούμε έτσι ώστε να βελτιωθεί. Δεν νομίζω λοιπόν ότι στο Συμβούλιο υπάρχουν κράτη-μέλη τα οποία θα χρησιμοποιήσουν το ε, νέο σύστημα επίλυσης διαφορών ε, για να μπλοκάρουν την ε, ολοκλήρωση της Συμφωνίας ΣΥΤΑ. Τώρα, ισχύει αυτό που είπατε ότι δεν έχουμε ολοκληρώσει πολλά, πολλά νομοθετικά έργα, όμως είναι δύσκολο και πρέπει, ξέρετε, να συμφωνήσουν όλα τα κράτη-μέλη για κάτι. Υπάρχουν κάποιες χώρες οι οποίες μπλοκάρουν τα πράγματα εδώ και πάρα πολύ καιρό και πιστεύω και εγώ πως είναι καιρός να σταματήσει αυτό. Ως Προεδρία όμως ε, σας διαβεβαιώ ότι κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να ε, υπάρχει ένα πνεύμα συνένεσης έτσι ώστε να προχωρήσουμε και στους ε, τιμερείς διαλόγους. Πολύ ωραία. Ε, Τζουν. Σας ευχαριστώ πολύ. Δύο σύντομες ερωτήσεις. Η πρώτη έχει να κάνει με τον Χάλιβα. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ότι ο κλάδος αυτός είναι πάρα πολύ σημαντικός για την Ευρώπη. Αποτελεί πραγματικά τη βάση της βιομηχανικής μεταποιητικής μας δραστηριότητας. Δεν ξέρω λοιπόν αν ο αποκλεισμό που είχε προβάλει το Μένο Βασίλειο είχε αρθεί αυτή τη στιγμή και αν συνεχίζονται οι διαπραγματεύσει στα πλαίσια του Συμβουλίου. Σε σχέση επίση με τον εξυγχρονισμό των μέσων αμυντικής άμυνας. Πέρα από αυτό, το Συμβούλιο προχωρά και σε άλλε διαπραγματεύσει προκειμένου να αντιμετωπίσει την κρίση στον τομέα του Χάλιβα. Δεύτερη τώρα ερώτηση, οι σχέσει μα με τι χώρε Αφρική και οι συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης. Ξέρετε ότι οι συμφωνίες αυτές έχουν ένα πολύ αδύναμο κεφάλαιο όσον αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη. Από τότε που ξεκίνησε μάλιστα και η Global Europe Agenda στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από ό,τι φαίνεται αποδυναμώνονται η δική μας στάση στα πλαίσια των συμφωνιών αυτών για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Έχει απασχολήσει αυτό το Συμβούλιο και αν έτοχετε ναι, ζητήσει ως επίγον ζήτημα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Bon, sur... Euh, Όσον αφορά το χάλιβα, δεν άλλαξε στάση το Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό το οποίο συζητήσαμε, και το λέω με απόλυτη σοβαρότητα, ήταν αν μπορούμε να κάνουμε ένα διαχωρισμό ανάμεσα στο χάλιβα και τα προβλήματά του και το καθεστώς οικονομίας της αγοράς για την Κίνα. Συζητήσαμε λοιπόν τα δύο αυτά ζητήματα. Όσον αφορά την αγνώριση του καθεστώτο οικονομία τη αγορά στην Κίνα, είναι τρει συναλλακτικέ. Ή δεν κάνουμε τίποτα απολύτω, ή αλλάζουμε τα πάντα, ή διαπραγματευόμαστε. Προκειμένου να καταλήξουμε δηλαδή σε μια συμφωνία με την Κίνα για κάποιου τομεί όπω ο Χάλιβα ή όπω τα φωτοβολταϊκά πάνελ κτλ. Αυτό απασχόλησε τα περισσότερα κράτη-μέλη και σε κάθε περίπτωση, όπως είπαμε για τον Χάλιβα, υπάρχουν 350 θέσεις απασχόλησης οι οποίες εξαρτώνται άμεσα από το τομέα του Χάλιβα, το διπλάσιο ενδεχομένω για τις έμεσες θέσεις απασχόλησης. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να δούμε τι γίνεται και αν το Ηνωμένο Βασίλειο προβλέπει από τώρα ότι θα υπάρχουν προβλήματα, ότι τα πράγματα είναι όντω σοβαρά. Η Ευρώπη λοιπόν θα πρέπει να παραμείνει ανοιχτή και διαλλακτική όσον αφορά τον τομέα του εμπορίου, αλλά για το συγκεκριμένο αυτό ζήτημα νομίζω ότι κατά τη διάρκεια της Ολλανδικής Προεδρίας και ενδεχομένως και κατά τη διάρκεια της Σλοβακικής Προεδρίας που θα ακολουθήσει και συμφωνεί με αυτό και η Επίτροπος είναι πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε το ζήτημα αυτό είναι πάρα πολύ ευαίσθητο. Γι' αυτό το λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει καταλήξει ακόμα σε οριστική απόφαση. Συνεχίζονται συζητήσει και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Συμβούλιο. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να, να δούμε πώ συνδέεται το ζήτημα αυτό τη Κίνα με τον κλάδο του Χάλιβα. Όσον αφορά τώρα την Αφρική. Θα κάνουμε κάθε τι το δυνατό έτσι ώστε μετά τη σύνοδο της Μάλτας, στην οποία έλαβα και εγώ μέρος, σύνοδος για τη μετανάστευση, φάνηκε η βούληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην αυξήσει απλώς και να εντείνει τις σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αφρικής όσον αφορά το ζήτημα της μετανάστευσης αποκλειστικά, ότι θα πρέπει να προσφέρουμε περισσότερα πράγματα στην Αφρικανική Ήπειρο. Στο πνεύμα λοιπόν αυτό και εσείς και εμείς στην Ευρωπαϊκή στο Συμβούλιο, με συγχωρείτε, μπορούμε να καταβάλουμε σημαντικές προσπάθειες για να ενισχυθεί η σχέση ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Αφρική. Σα um, Σας ευχαριστώ. Ακούστηκαν πολλά, δεν θα θέσω πολλές ερωτήσεις. Θέλω να ακούσω όμως για τα ορυκτά προϊόντα περιοχών συγκρούσεων. Μπορείτε να μας πείτε πού βρισκόμαστε και πότε μπορούμε να περιμένουμε μια συμφωνία και ποια είναι τα τελευταία εμπόδια τα οποία αντιμετωπίζουμε από κάποιες χώρες. Πολύ θα θέλαμε να ξέρουμε ποιοι τα βάζουν. Μπορώ να μιλήσω γερμανικά μαζί σας. Λοιπόν, δεν γνωρίζω αν πρέπει να ονομάσω συγκεκριμένες χώρες, αλλά να σας πω ότι υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά το ποιος είναι η αρμόδια αρχή. Πιστεύω όμως ότι Είναι θέμα πολιτικής. Και σίγουρα χρειάζεται και οφείλουμε να βρούμε κάποια συνένεση μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι ώστε τα προϊόντα που εισάγουμε να μην προέρχονται από περιοχές όπου λαμβάνουν χώρα συγκρούσεις μπορεί να αρχίσει ο τριμερής διάλογος από το Συμβούλιο. Εμείς δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα και από ό,τι γνωρίζω ο τριμερής διάλογος θα αρχίσει κατά τη διάρκεια της δικής μας προεδρίας. Είναι δύσκολο. Μ, λίγο δύσκολο, μου λέει ο συνάδελφος. Είμαστε μία μικρή χώρα. Ε, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον Υπουργό για την πληρέστατη παρουσίαση για τις διαπραγματεύσεις με την Τίνιδα. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να γνωρίζουμε περισσότερα. Θα ήθελα επίσης να ληφθεί υπόψη η συμφωνία ε, στην οποία έχουμε καταλήξει για το ελαιόλαδο και πόσο θα μπορούσε αυτή η συμφωνία να επηρεάσει κάποιες ε, περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει μια τέτοια μελέτη στην Ιταλία, στην Ισπανία, την Πορτογαλία και την Ελλάδα. Έτσι και αλλιώ μια τέτοια συμφωνία, έστω και για ένα χρόνο, μετά το χρόνο θα πρέπει να δούμε τα αποτελέσματα που θα προκαλέσει σε αυτές τις περιφέρειες και τότε να αποφασιστεί αν θα παραταθεί για ένα επόμενο. Ναι, αυτή είναι η τελευταία απάντηση που μπορώ να δώσω. Έχω ένα διαδικαστικό σημείο, κύριε Πρόεδρε. Υπάρχει... Υπάρχει μεγάλη ανησυχία για μας για τις διαδικασίες. Η διαδικασία λοιπόν την οποία θέλω να ρωτήσω στον κύριο εκπρόσωπο του Συμβουλίου και δεν θα τα καταφέρω. Και εξαρτώμαι από την καλή βούληση του Υπουργού να μου επιτρέψει να θέσω ένα ερώτημα το οποίο είχα δικαίωμα να θέσω έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, για το ελαιόλαδο καταρχάς. Ο Πρωθυπουργό της Τινησίας είχε έρθει στο Συμβούλιο, συζητήσαμε μαζί του το θέμα αυτό και με τις χώρες οι οποίες ενδιαφέρονται ιδιαίτερα που είναι ελαιοπαραγωγή, το μέτρο είναι προσωρινό και το Συμβούλιο ομόφωνα είπε ότι βρίσκεστε σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση, πρέπει να σας βοηθήσουμε χωρίς να κάνουμε στην παρούσα φάση αν θέλετε ε, προβλέψεις για πιθανές ζημίες σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι 28 χώρες αφού άκουσαν τον Πρωθυπουργό της Τινησίας πήραμε αυτή την απόφαση και δόθηκαν εγγυήσεις στις χώρες παραγωγής ότι το μέτρο αυτό είναι αυστηρά προσωρινό. Ευχαριστώ Υπουργέ, ο κύριος Ντάτμουθ και κύριοι συνάδελφοι σας εγγυώμαι ότι αν δώσετε μία γραπτή ερώτηση θα τη μεταφέρω στον κύριο Άσελμπορν και θα δώσει τις απαιτούμενες απαντήσεις. Και αν δεν απαντήσει θα τον πιέσω πάρα πολύ να το κάνει αυτό έτσι ώστε όλοι να μπορέσουν να εκφραστούν. Γιατί αλλιώς ε, φοβάμαι ότι θα αδικήσουμε τα μέλη του Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ όλους που μας δώσατε μια συνολική παρουσίαση και θα στείλουμε την ομιλία σας σε όλους. Διαδικαστικό, αφού φύγει ο Υπουργός Άσεμπον, έχω ένα διαδικαστικό, λέω Λοβδοτάκμου. Is this the final? it's not Κύριε Πρόεδρε, διαδικαστικό. Πολύ ευγενικό εκ μέρου σα να δεχθείτε γραπτέ ερωτήσει όπω είπατε. Αλλά και εσεί είστε ευρωβουλευτή πολύ περισσότερο από μένα. Ξέρετε ότι χρειάζονται 5-6 εβδομάδε για να καλυφθούν αυτέ οι γραπτέ ερωτήσει. Επομένω, δεν νομίζω ότι είναι αποτελεσματικό το σύστημα αυτό. Θα μπορούσαμε να καθορίσουμε μια συγκεκριμένη διαδικασία. Η διαδικασία καταρχά είναι ότι ακούμε πρώτα του συντονιστέ. Έτσι δεν είναι. Εσείς άλλο δρόμο ακολουθήστε εδώ πέρα. Ο κύριος Φίσας Αγέλα έθεσε ένα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα, αλλά είπατε ξαφνικά ότι ήταν το τελευταίο ερώτημα το οποίο μπορούσατε να δεχθείτε, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι η δική μου πολιτική ομάδα δεν ακούστηκε καθόλου σε αυτή τη συζήτηση. Η διαδικασία κανονικά είναι ότι Ακούγουμε πρώτα τους συντονιστές των πολιτικών ομάδων. Δύο φορές ακούσαμε μιλητέ από το ΕΛΚ, Καμία φορά δεν πήραμε εμεί το λόγο. Ποια είναι λοιπόν ακριβώ τη διαδικασία. Ακολουθείτε μια άλλη διαδικασία σα από σήμερα. Τι ακριβώ συμβαίνει. Καταρχά σα εγγυώμαι ότι ήδη μέχρι τα τέλη του έτου θα έχετε λάβει μια απάντηση. Και δεύτερον, ακόμα και οι ευρωβουλευτέ από του φιλελεύθερου και την ΚΟΕ δεν κατάφεραν να πάρουν το λόγο. Δεν είστε μόνο εσεί. Και αυτό επειδή πιέζει ο χρόνο. Ξέρω ότι τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Επικράτησε μια κάποια σύγχυση. Δεν μπορούσα βέβαια να κάνω τον Υπουργό να μείνει περισσότερο. Ναι, αλλά αν πρόκειται για κάποιο νέο κανόνα, εμείς θα την εγκρίναμε. Εγώ είχα απλώ μπροστά μου τον κατάλογο των ανθρώπων που είπαν ότι θέλουν να πάρουν το λόγο, που σήκωσαν το χέρι προτού ξεκινήσει η συζήτηση. Αυτό συνέβη. Πολύ ωραία. Περνάμε λοιπόν στο σημείο 18. Τα επόμενα δύο σημεία της ημερήσιας διάταξης είναι θέματα τα οποία μπλοκάρονται από το Συμβούλιο. Το 18 έχει να κάνει με την IPI, στο οποίο αναφέρθηκε ο Υπουργός. Τον Ιανουάριο του 2014 εγκρίθηκε από εμάς, ήταν η έκθεση Κασπάρη. Και τώρα μένει να δούμε τι θα κάνουμε έτσι ώστε να υπάρξει πρόοδος. Θα δώσω τώρα το λόγο στον εισηγητή Ντάνιελ Κασπάρη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αναφερθήκατε ήδη στα ουσιώδη. Εμείς κάναμε τη δουλειά μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αυτό που θέλουμε είναι να μην ξεχαστεί αυτό το θέμα. Ψηφίστηκε στο Κοινοβούλιο και το ευκταίο θα ήταν εάν καταφέρνα να συμφωνήσουν το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι ώστε να ε, προχωρήσουμε. Πώς μπορούμε λοιπόν να κινήσουμε τα πράγματα. Ε, ευχαριστώ. Υπάρχουν σχόλια από τους συναδέλφους. Δεν βλέπω σχόλια. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το IPI. Ποιος θα ήθελε να μιλήσει. Ο κύριος Γέσεν. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πολύ σύντομα να σας πω ότι αυτή η πρόταση υποβλήθηκε από κοινού το 2014 και στόχος ήταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποκτήσει μεγαλύτερη μόχλευση με τους εμπορικούς εταίρους έτσι ώστε οι Ευρωπαίοι προμηθευτές να μπορούν να ε, λαμβάνουν μέρος σε διαγωνισμούς για δημόσιες ε, συμβάσεις σε τρίτες χώρες. Έχω μελετήσει τον φάκελο πολύ προσεκτικά και προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να εισέλθουμε σε διαβουλεύσεις με τους κύριους ενδιαφερόμενους φωνείς και τα κράτη-μέλη. Σήμερα μπορούμε να ανακοινώσουμε ότι γίνεται μία ε, διυπηρεσιακή διαβούλευση έτσι ώστε να ε, ε, δημοσιευτεί μία νέα πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον Ιανουάριο. Άρα λοιπόν προχωρά το θέμα μπορώ να σας πω. Μάλιστα, τον Ιανουάριο λοιπόν θα κοινοποιηθεί μία αναθεωρημένη και επικαιροποιημένη πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βρίσκεται κάποιος εκπρόσωπος του Συμβουλίου εδώ. Όχι. Τάνιελ, θέλει να προσθέσεις κάτι, να σχολιάσεις. Ωραία. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα γίνει τον Ιανουάριο. Ναι, έρχονται Χριστούγεννα, πολλές εκπλήξεις θα έχουμε να δούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να δούμε τι θα μας αφήσει λοιπόν στο δέντρο. Περνάμε στο σημείο 19. TDI και εδώ μπλοκάρει το Συμβούλιο. Τον Απρίλιο του 2014 αποφασίσαμε ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα και είναι καιρός να προχωρήσουμε έτσι ώστε να δρομολογήσουμε τον εξυγχρονισμό του TDI. Ο κ. Χέλνερ είναι υπεύθυνο και έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Άκουσα με μεγάλο ενδιαφέρον τον Υπουργό του Λουξεμβούργου που αναφέρθηκε σε αυτό, σε αυτήν την έλλειψη δυστυχώς πρόοδου. Θα ήθελα ε, όμως ε, να πω επίσης ότι όπως αναφέρετε και εσείς ε, το θέμα αυτό συζητιέται και στα πλαίσια της πρόσβασης στην αγορά της Κίνας και την ε, ανακήρυξη της οικονομία της αγοράς. Το θέμα όμως δεν είναι πιστεύω αυτό, το θέμα είναι τα ε, μέσα που έχουμε έτσι ώστε να... τα αμυντικά εμπορικά μέσα μάλλον που διαθέτουμε. και το πώς θα προχωρήσουμε. Θα ήθελα λοιπόν να μάθω και την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διότι έγινε η συνεδρίαση και κλεισμένων των θυρών με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όμως δεν έχουμε ακούσει νεότερα σχετικά με το πώς συνδέονται αυτά τα θέματα. Εγώ προσωπικά θα ήθελα να πω ότι το θέμα της οικονομίας της αγοράς, το χαρακτηρισμού αυτού για την Κίνα, δείχνει τις αδυναμίες στην πρόταση της Επιτροπής. Δεν αναφέρθηκε καν αυτό το καθεστώς οικονομίας της αγοράς στην πρόταση της Κομισιόν. Γι' αυτό λοιπόν ως συνέπεια αυτού απορρέει το τι θα, τι θα κάνουμε, πώς θα αντιδράσουμε και είναι πάρα πολύ σημαντικό επίσης και το θέμα των επιχορηγήσεων. το οποίο επίσης δεν συζητήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεν αναφέρθηκε στην πρόταση της Επιτροπής. Θα ήθελα λοιπόν να μάθω τι άποψη έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γι' αυτό. Και τέλος, να σημειώσω ότι αυτή η πολύ ισορροπημένη συμβιβαστική πρόταση στην οποία καταλήξαμε στο Κοινοβούλιο δεν έχει ε, οδηγήσει σε συζητήσεις στο Συμβούλιο για το καθεστώ και, και της Κίνας. Και θα ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει κάποια διαφορά. Ευχαριστώ πολύ. Το θέμα είναι η διαφάνεια. Υπάρχει ο κατάλογος εδώ, κυρία Μόσκα, κύριο Μπορέλη, κύριο Τάρτμαουθ, κυρία Ροντρίγκεφ και η κυρία Ρέντινγκ. Και η Αμαμαρ Κλάγκλιν θα λάβουν το λόγο. Σας παρακαλώ να είστε σύντομοι. Δεν θέλω να επαναλάβω πράγματα, θα ακολουθήσω αυτά τα οποία υπεθύμησε ο προηγούμενος συνάδελφος. Επανειλημμένα έχουμε εκφράσει τη δυσφορία μας ε, για το ότι έχει παγώσει το σημαντικό αυτό θέμα. Να πω ότι με ανασύχησε σε σχέση με αυτά τα οποία άκουσα από τον εκπρόσωπο της Προεδρίας του Λουξεμβούργου την δυνατότητα η οποία φαίνεται ότι μελετάτε να υπάρξει μια διαρρύθμιση σε σχέση με την διάσωση ορισμένων τομέων, μια δηλαδή προσπάθεια να δοθεί προτεραιότητα σε ορισμένους τομείς εις βάρος κάποιων άλλων. Κάτι το οποίο θα επιβαρύνει τις συνέπειες σε συγκεκριμένους τομείς και όχι τόσο σε κάποιους άλλους. Θα ήθελα να μάθω λοιπόν να έχω κάποιες διευκρινήσεις πάνω σε αυτό γιατί η πολυδιάσπαση ανατομέα δεν είναι μια γραμμή στην οποία συμφωνούμε. Ο κύριος Μπορέλη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η ανάγκη εξυγχρονισμού των μέσων άμυνας επιθετικών και ε, των μέσων άμυνας των συμπερόντων εννοώ είναι κάτι το πάρα πολύ θετικό. Νομίζω ότι η προσπάθεια που κάναμε ήταν ε, οδήγησε σε ένα ισορροπημένο κείμενο το οποίο αποδέχεται το επιχειρηματικό και παραγωγικό μας σύστημα. Δεν θα πρέπει να το υπονομεύσουμε αυτό. Έγινε πολύ καλή δουλειά λοιπόν στο Κοινοβούλιο η οποία έχει μπλοκαριστεί τώρα στο Συμβούλιο για διάφορους λόγους διαφοράς στις εθνικές θέσεις. Θα ήθελα να περιοριστώ λοιπόν εγώ στην ανάγκη να σεβαστούμε το κείμενο, να εμείνουμε στο κείμενο το οποίο είχαμε διατυπώσει εδώ για δύο, για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί είμαι πεπισμένος ότι οι θέσεις του Κοινοβουλίου είναι και σήμερα σωστές και νομικά και πολιτικά και οικονομικά. Δεύτερον, είναι προφανές ότι με το πέρασμα του χρόνου είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπάρξει ενημέρωση της οδηγίας αυτής λόγω της δυναμικής της αγοράς και θα ήθελα επίσης να θέσω κάποια θέματα τα οποία θεωρώ κρίσιμα για τη συζήτησή μας. Τα μέσα ε, εμπορικής άμυνας αν θέλετε έχουν μεγάλη σημασία για την προστασία των επιχειρήσεών μας στρεβλές εμπορικές πρακτικές. Τα μέσα αυτά θα μας επιτρέψουν να ενισχύσουμε την προστασία των επιχειρήσεων και αυτό είναι καλό. Αυτό σημαίνει λιγότερος χρόνος εξέτασης και όχι εννέα μήνες. Διαπίστωση του ντάμπινγκ δεν απαιτεί τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Ποτέ δεν μπορούμε να είμαστε, θα έλεγα, εύθετοι στο χρόνο μας. Καλό θα είναι το εννέα μήνες να γίνει επτά Τώρα για τον λεγόμενο προβλεπτό κίνδυνο ή κίνδυνο ζημίας καλύτερα και εδώ είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αξιολογηθεί σωστά. Ένα άλλο θέμα είναι η διατύπωση κανόνων πολύ πιο εύκολα ερμηνεύσιμων για την καταγραφή των εξαγωγικών προϊόντων πριν από την πραγματική εξαγωγή. Αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ τις μικρομεσές ε, και νομίζω ότι θα δεις γλιτώσει πολλές γραφειοκρατικές διαδικασίες. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Οι περισσότεροι το ξέρουμε και η κυρία Κέρτον Ντάρλινγκ το είπε επίση ότι στον τομέα του Χάλιβα στη χώρα μου βρισκόμαστε σε έκτακτη κατάσταση. Έγραψα στις 22 Οκτωβρίου στον, στην Επίτροπο ζητώντας να υπάρχουν μέτρα για τις εισαγωγές προϊόντων χάλιβα από την Κίνα προς το Μέντο Βασίλειο. Μόλις χθες έλαβα την απάντηση, η οποία μεταξύ άλλων λέει ότι δεν μπορούν να επιβληθούν μέτρα αντι-dumping χωρίς να καθορίζουμε πρώτα ότι όντως λαμβάνει η χώρα dumping ή επιδότηση στις παρατηρήσεις του, ο Υπουργός από το Λουξεμβούργο είπε ότι έχουμε αθέμητο ανταγωνισμό. Αυτό τι σημαίνει στην πράξη, dumping σημαίνει. Άκουγα βέβαια την διερμηνία, έχουμε μεταφρασμένο το κείμενο. Πιστεύω πάντως ότι θα πρέπει να διανεμηθούν τα πρακτικά ουσιαστικά. Και όσον αφορά το Χάλιβα, και το ξέρετε πολύ καλά πρόεδρε, όταν πραγματικά οι κλίβανοι ουσιαστικά σταματά να λειτουργούν, δεν μπορούν στη συνέχεια να επανέλθουν σε κατάσταση λειτουργίας. Και αυτό που έχουμε δει τώρα είναι ότι η Επίτροπος για το Εμπόριο, σε συνεργασία με το Συμβούλιο, αντιμετωπίζει αυτή την επίγουσα κατάσταση με μια στάση γραφειοκρατική, νοχελική, σε κατάσταση λιθάργου θα έλεγα. Πιστεύω λοιπόν ότι ή θα συμβεί τίποτα ή αυτό θα πετήσει πάρα πολύ χρόνο. Καταλαβαίνετε όμως ότι επιτόπου για τη βιομηχανία θα είναι πάρα πολύ αργά. Δεν νομίζω ότι θα έπρεπε εγώ να είμαι μονομένο και μόνος μου να κάνω την έκκληση αυτή. Απευθύνομαι τώρα στους συναδέλφους μου. Καλό λοιπόν τους συναδέλφου να μου υποστηρίξουν για το ζήτημα αυτό, προκειμένου να θέσουμε εκ νέου το ζήτημα αυτό και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Συμβούλιο. Εγώ θα πρότεινα ότι δεν θα έπρεπε καν να απευθυνθούμε βέβαια σε αυτό σε αυτούς τους δύο οργανισμούς. Αναγκαστικά όμως πρέπει να το κάνουμε, να κάνουμε μια έκκληση προκειμένου να έχουμε επίγοντα μέτρα από το Συμβούλιο και την Επιτροπή προτού να είναι πολύ αργά. Ευχαριστούμε πολύ, Μάρα. Ευχαριστώ. Αυτό το οποίο θα ήθελα να πω είναι ότι λυπάμαι αυτό το οποίο συνέβη με τον κύριο Άσεμποργκ γιατί μένα με ανησύχησαν αυτά τα οποία είπε. Ε, δεν μου απέδειξε ότι κατανοεί ε, θα έλεγα ε, την ανάγκη που υπάρχει και τον κατεπίγοντα χαρακτήρα εξυγχρονισμού των μέσων για την άμυνα των εμπορικών συμφερόντων. Πάρα πολλοί τομεί θίγονται γιατί δεν υπάρχει σεβασμός των κανόνων από τον πλευρά του ανταγωνισμού σε συνδυασμό και με τους ε, περιορισμούς για την προστασία του περιβάλλοντος και το υψηλό κόστος της ενέργειας, ο ανταγωνισμός δεν είναι δίκαιος. Δεν μπορούμε λοιπόν παρά να εξυγχρονίσουμε τα μέσα εμπορικής άμυνας και ξέρουμε τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν όταν εξαφανιστεί ή δεν γίνει πλέον σεβαστό και δεν εφαρμόζεται το άρθρο 15. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε λοιπόν να πείσουμε τα κράτη-μέλη, θα πρέπει να το συζητήσουμε το θέμα αυτό και σε εθνικό επίπεδο, γιατί δεν μπορεί να περιμένει άλλο τους χρόνους ε, λειτουργίας και αναθεώρησης του Συμβουλίου. Ε, υποτίθεται ότι είμαστε υπέρ της επαναβιομηχάνησης ενώ ε, την ίδια στιγμή αφήνουμε τις βιομηχανίες, τις ανταγωνιστικές να βυθίζονται. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο Υπουργός του Λουξεμβούργου, αν είχε παραμείνει λίγο εδώ, θα ήθελα να του θέσω παρουσίαν του αυτό το ερώτημα, γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Όσον αφορά την εμπορική άμυνα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέλαβε δράση, το ίδιο έκανε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το ίδιο έκανε και μάλλον τώρα μπλοκάρει το Συμβούλιο. Και Μαθαίνουμε από την Λουξεμβουργιανή Προεδρία ότι προσπάθησε να ξεμπλοκάρει την κατάσταση και μας είπε ότι συζητάνε με τους υπουργούς για τα σημαντικά προβλήματα της χαλιβουργίας, αλλά ότι από την άλλη δεν αναλαμβάνεται δράση προκειμένου να εγκρίνουμε κάποιο μέσο εμπορικής άμυνας. Και ουσιαστικά δεν λέμε τίποτα συγκεκριμένο όσον αφορά το καθεστώς οικονομίας αγοράς για την Κίνα και το τι γίνεται με τις αγωγές πρώτων χάλιβα και αυτή τη στιγμή Πραγματικά δεν γνωρίζουμε ποιο συζητεί με ποιον και για ποιο ζήτημα. Δεν μπορώ να καταλάβω ποια είναι η λογική που ακολουθείτε. Έχουμε μπροστά μα ένα συγκεκριμένο σοβαρό πρόβλημα. Πρέπει να λάβουμε σοβαρέ αποφάσει και από ό,τι φαίνεται το Συμβούλιο δεν κινείται καθόλου αυτή τη στιγμή. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Ευχαριστούμε πολύ, Έμα. Κοιτάξτε, είναι σαφές ότι ε, τα μέσα εμπορικής άμυνας πρέπει να επικαιροποιηθούν. Αυτά που χρησιμοποιεί δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο πρέπει να κάνει το συντομότερο δυνατό τις αλλαγές αυτές. Για ποιο λόγο μας ανησυχεί τόσο πολύ η κατάσταση αυτή με τα μέσα εμπορικής άμυνας. Υποτίθεται ότι τα μέσα αυτά θα πρέπει να προστατεύουν από τον αθέμητο ανταγωνισμό την, εμπορική, την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για τον τομέα της χαλιβουργίας. Έχουμε πάρα πολλέ εισαγωγές προϊόντων χάλιβα από την Κίνα με τιμές πάρα πολύ χαμηλές, σε πολύ χαμηλότερες από αυτές που έχουμε σε χώριο επίπεδο. Άρα μιλάμε για dumping. Για ποιο λόγο λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν κάνει κάτι, πώς παρακολουθεί την κατάσταση όσον αφορά τα μέσα εμπορικής άμυνας και πώς παρακολουθεί τις σχέσεις τις εμπορικές που έχουμε με τρίτες χώρες. Πόσο στενά παρακολουθεί λοιπόν την κατάσταση και τι κάνει για τις χώρες που πλήττονται και τι προτίθεται να κάνει στο μέλλον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να λάβει μια προληπτική δράση στο μέλλον και να έχει και ένα σύστημα έγκαιρη προειδοποίηση προκειμένου να μπορούμε πολύ γρήγορα να λαμβάνουμε δράση και να αποφεύγουμε κάθε αθέμητη εμπορική πρακτική όπω τώρα με την περίπτωση αυτή dumping, έτσι ώστε να μην πλήττονται οι ευρωπαϊκέ βιομηχανίε. Τελειώνει ο χρόνο, δεν μπορούμε να ακούμε πλέον δικαιολογίε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θέλουμε συγκεκριμένα μέτρα. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα ο Φρανκ θα έχει την ευκαιρία να απαντήσει σε αυτές τις ερωτήσεις. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητά κύριε Λάνια. Θα ήθελα καταρχάς να κάνω μια σύντομη δήλωση σχετικά με την κατάσταση του θέματος του εξυγχρονισμού και μετά επιτρέψτε μου να κάνω ορισμένα σχόλια και κάποια εκτιμήσει σχετικά με αυτά που είπαν οι ευρωβουλευτέ. Ο κ. Σεφίλνε μα είπε ότι η πρόταση είναι από τον Απριλίο του 2013, ότι έχει συζητηθεί εκτενέστατα εδώ και πώς η πρώτη έγκριση έλαβε χώρα τον Απρίλιο του 2014. Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουμε παρατηρήσει ότι το Συμβούλιο έχει προσπαθήσει να ε, δρομολογήσει το θέμα. Η Ιταλική Προεδρία μάλιστα είχε καταβάλει έντονες προσπάθειες και επίσης είχε κάποιες ε, συγκεκριμένες προτάσεις. Είχε ε, κυκλοφορήσει ένα κείμενο στην ομάδα εργασίας, δεν κατάφερε όμως να προχωρήσει παραπέρα. Φέτος το 2015 η Λετωνική Προεδρία θεωρούμε πως δεν ήταν ιδιαίτερα δραστήρια. Η Προεδρία του Λουξεμβούργου ε, προσπάθησε να σκεφτεί το που βρίσκονταν τα κράτη-μέλη σχετικά με την πρόοδο του θέματος, όμως ε, δεν κατάφερε να ε, φτάσει σε κάποια συνένεση. Έτσι λοιπόν δεν, ε, δεν καταφέραμε να προχωρήσουμε. Γι' αυτό λοιπόν δεν νομίζω πως η Προεδρία του Λουξεμβούργου θα πάει το θέμα παραπέρα. Τώρα, από ό,τι καταλαβαίνω, στο Συμβούλιο υπάρχει γενική αίσθηση πως υπάρχει ο συνήθις διχασμός ανάμεσα στα κράτη-μέλη, ανάμεσα σε εκείνα που από τη μία είναι περισσότερο υπέρ της προστασίας της βιομηχανίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της παραγωγής της Ένωσης και από την άλλη υπάρχουν τα κράτη-μέλη εκείνα όπου ε, είναι υπέρ του ελεύθερου εμπορίου και των προϊόντων από, τρίτες, ε, από τρίτους ε, προμηθευτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει λοιπόν αυτή η βασική ε, διαφωνία, όμως να σας πω ότι στο Συμβούλιο υπάρχουν αρκετές αντιπροσωπείες οι οποίες θεωρούν πως η θέση του Κοινοβουλίου δεν είναι αρκετά ισορροπημένη. Και αυτό συνεισφέρει στο μπλοκάρισμα που αναφέρεται. Τώρα, ο κύριος Φιέλνερ δεν μας ε, με βρίσκει μη σύμφωνο όσον αφορά τις ε, επιδοτήσεις των κρατών μελών. Πιστεύω πως ε, δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε τον κανόνα των μικρότερων δασμών σε τις περιπτώσεις επιδοτήσεων. Και αυτό το παρατηρούμε σε ορισμένες περιπτώσεις πολύ μεγάλων επιδοτήσεων που οδηγούν σε αθέμητο ανταγωνισμό. Χρειάζεται λοιπόν εξυγχρονισμός, αλλά πολύ σωστά είπε ότι σίγουρα το 2013 βρισκόμασταν ακόμα σε πρώιμο στάδιο της Τώρα, ίσως ακούσατε όλοι σήμερα νωρίτερα πως ο κύριος Άσελμπορν είπε ότι αναμένουμε τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο MES για την, και να, πως πρέπει να προσπαθήσουμε να επηρεάσουμε τα κράτη-μέλη έτσι ώστε να προχωρήσουν σε αυτόν τον εξυγχρονισμό. Έτσι λοιπόν καταλαβαίνω εγώ τα πράγματα ότι η Προεδρία της Ολλανδίας θα περιμένει τη θέση των κρατών μελών για το καθεστώς οικονομίας της αγοράς και θα προσπαθήσει να βρει την κατάλληλη ισορροπία έτσι ώστε να προστατεύσει την ευρωπαϊκή βιομηχανία και σύντομα και από την άλλη να μην ε, σαμποτάρει τον ίδιο της ε, τον εαυτό μειώνοντας ε, τον όγκο του νόμιμου εμπορίου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν θα βοηθήσει όσο μπορεί την Ολλανδική Προεδρία. Εμείς θα δώσουμε τη στήριξή μας στις μελλοντικέ συζητήσεις. Προς το παρόν όμως πρέπει να σας πω πως δεν νομίζω να γίνει αυτό ε, τώρα μέχρι το τέλος της Προεδρίας του ε, Λουξεμβούργου και να φτάσουμε σε κάποια συγκεκριμένη θέση για το καθεστώς οικονομίας της αγοράς. Τώρα, σχετικά με τις ε, παρεμβάσεις κάποιων ευρωβουλευτών, να σας πω πως, ναι, επί της ουσίας συμφωνώ και συμφωνούμε πως χρειάζεται μια γρήγορη και αποτελεσματική διεκπαιρέωση των ε, διάφορων εφακέλων, όμως καταρχάς βλέπουμε πως υπάρχει, υπάρχουν αντιδράσεις, υπάρχουν ενστάσεις από την ε, ίδια την αγορά για τις περιπτώσεις ε, dumping. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν πρέπει να δημιουργήσει τον βασικό κανονισμό και επειδή μας διέπουν κανόνες ακριβώς δεν μπορώ να σας πω ότι μπορούμε να δράσουμε έτσι αυθαίρετα. Χρειάζεται να γίνουν κάποιες αναφορές, να γίνουν κάποιες ενστάσεις. Και τότε, σε αυτήν την περίπτωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάντα προσπαθεί να λύσει τα προβλήματα που προκύπτουν και να επιταχύνει την διαδικασία αυτή. Να είστε σίγουροι ότι αυτό το θέμα είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό και έτσι το αντιμετωπίζουμε. Επίσης, νομίζω κάποιος άλλος ευρωβουλευτής είπε πως είναι πολύ δύσκολο να αντιδράσουμε σε περίπτωση κάποιας απειλής παρά σε περίπτωση που ήδη διαπιστωθεί ε, πως ε, συμβαίνει αυτό το dumping. Υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες, πρέπει να σας πω, και εάν έχουμε κάποια τέτοια καταγγελία, τότε ε, δρούμε. Τώρα, κύριε Ρέντινγκ, Είπατε πως πράγματι δεν υπάρχει συμφωνία ανάμεσα στους υπουργούς στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητα σχετικά με τον Χάλιβα και σε εκείνους του Συμβουλίου Εμπορίου που υποστηρίζουν πόσο ε, ο πρέπει να γίνει στο σωστό χρόνο. Μην ξεχνάμε πως πρέπει και τα κρατημέλη να κάνουν πρόοδο έτσι ώστε να καταφέρουμε να συγχρονιστούμε όλοι. Και εδώ, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ολοκληρώσω τα σχόλιά μου για ε, αυτά που ακούσαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Υπάρχουν κάποια σχόλια παραπάνω. Ευχαριστώ πολύ. Να σας πενθυμίσω δύο πράγματα όσον αφορά το ζήτημα της χαλιβουργίας που μας απασχολεί όλους. Πολύ πρόσφατα, πριν από ένα μήνα, πριν από μερικές εβδομάδες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε την ε, έκδοση των τελευταίων αριθμητικών δεδομένων όσον αφορά τι εισαγωγέ προϊόντων χάλιβα. Εκεί, και το λέω αυτό στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπάρχουν συγκεκριμένε αποδείξει όσον αφορά το dumping και τη ζημία. Καταλαβαίνω πάντως τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν επιμένει ότι ε, θα πρέπει να προχωρήσουμε περισσότερο με την αναγνώριση καθεστώτος οικονομίας αγοράς για την Κίνα αλλά δεν μπορούμε πραγματικά να λέμε ότι ε, την πρώτη φορά που έγινε η απόπειρα μεταρρύθμισης των μέσων εμπορικής άμυνας το 2013, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τότε, το 2013, μας είχε πει ότι ήταν πολύ πρόημο. Τώρα όμως πλέον, το 2015, η κατάσταση είναι επίγουσα. Κάτι το οποίο ήταν πρόημο το 2013, ξαφνικά έχει γίνει έκτακτη ανάγκη το 2015. Συντοπίω επίσης ότι προφανώς έγιναν τροποποιήσεις όσον αφορά τους περιοριστικούς κανόνες για το anti-dumping, αλλά αυτό έγινε για όλα τα μέσα εμπορικής άμυνας και για τις επιδοτήσεις δηλαδή. Το θέμα τώρα είναι ότι αν η Κίνα πάρει το καθεστώς οικονομίας της αγοράς, θα πρέπει να γνωρίζουμε πώς ακριβώς θα συμβεί αυτό, με δική μας απόφαση, με απόφαση του ΠΟΕ, ανατομέα, συνολικά. Σε κάθε περίπτωση το ζήτημα αυτό των ε, μέσων εμπορικής άμυνας γίνεται αποδυναμώνεται ουσιαστικά κατά κάποιο τρόπο, γιατί για πάρα πολλά προϊόντα πλέον και για πάρα πολλού τομεί μπορεί μαζικά, συλλογικά να έχουμε εισαγωγέ που αποτελούν αντικείμενο dumping ή επιδοτήσεων. Νομίζω ότι αυτό το ζήτημα θα έπρεπε να μα απασχολήσει συλλογικά. Νομίζω ότι όπως είπε και ο εισηγητή, θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τους βασικούς κανονισμούς αντιντάμπινγκ και με το βασικό κανονισμό κατά των επιδοτήσεων. Αυτή τη στιγμή υπάρχει όμως μία πλειοψηφία στο Συμβούλιο Κρατών που μπλοκάρει την όλη διαδικασία. Συνεπώς, αν θέλουμε να καταλήξουμε σε θετικά συμπεράσματα, θα πρέπει και εμείς να πραγματευτούμε με το Συμβούλιο. Και μάλλον οι συνάδελφοι θα πρέπει να προετοιμαστούν για κάτι τέτοιο. Εκτενέστατα συζητήσαμε το ζήτημα αυτό το 2014 και τώρα βλέπουμε ότι μιλάμε για έναν πόλεμο τον οποίο καλούμεθα να νικήσουμε. Μέχρι στιγμής νικούσαμε μάχη ας μην χάσουμε όμως τώρα τον πόλεμο. Σίγουρα αυτό το είπα και πιο πριν εξάλλου στο TPC, Και Σιγητά, ότι το Κοινοβούλιο είναι ευέλικτο στις διαπραγματεύσεις του, όμως το πρόβλημα φυσικά είναι ότι το Συμβούλιο δεν έχει ακόμα εντολή για να εισέλθει σε διαπραγματεύσεις. Γι' αυτό λοιπόν ναι, είναι απόλυτα σαφές ότι το Συμβούλιο δεν βρίσκεται σε αυτό το στάδιο ακόμα. Όμως εμείς έχουμε μία εντολή και πρέπει να τη χρησιμοποιήσουμε. Και πρέπει σίγουρα να προσπαθήσουμε να βρούμε μία πιο ευέλικτη λύση. Περνάμε τώρα στο σημείο 20, ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Η Γεωγραφική ένδειξη είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Αύριο έχουμε την ολοκλήρωση της συμφωνίας με το ε, Βιετνάμ, όπου θα αναγνωριστούν 69 τέτοιες ονομασίες ε, γεωγραφικής προέλευσης. Και από την άλλη, βρισκόμαστε σε στάδιο διαπραγματεύσεων για τη συμφωνία TTIP και από ό,τι φαίνεται η αμερικανική πλευρά δεν έχει καμία πρόθεση να αναγνωρίσει το σύστημα αυτό. Υπάρχει λοιπόν όπως βλέπετε ένα τεράστιο εύρος απόψεων. Έχουμε καλέσει εδώ εμπειρογνώμονες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε εκπρόσωπο της ΓΔΑ Άγκρι, ο κύριος Κλάρκ, ο οποίος έχει έρθει συχνά στην Επιτροπή μας και με άλλη ιδιότητα. Σήμερα έχει έρθει για να μας παρουσιάσει την κατάσταση των πραγμάτων στις διαπραγματεύσεις σχετικά με τις ε, με τις γεωγραφικές ενδείξεις. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ο συνάδελφος Γένσεν, ο οποίος είναι διευθυντής στον τομέα του εμπορίου αγροτικών προϊόντων. Ευχαριστώ Τζον, ευχαριστώ και Πρόεδρε, με χαρά συμμετέχω σε μία θα έλεγα παρουσία εδώ. Έχουμε δύο συναδέλφους γιατί έχουμε μεικτή αρμοδιότητα και εγώ θα θέσω το γενικό πλαίσιο και ο Τζον Κλάρκ θα ασχοληθεί περισσότερο με λεπτομέρειες. Πρώτον θα ήθελα να πω ότι το σύστημα GI είναι μια προτεραιότητα που περιλαμβάνεται στο σωστό μέγεθος στην διεθνή μας εμπορική δραστηριότητα είναι κάτι το οποίο προσπαθούμε να ορίσουμε σωστά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά κυρίως φυσικά στις υποανάπτυξη χώρες και τις χώρες εμπορικούς εταίρους. Έχουν αλλάξει τα πράγματα τα τελευταία χρόνια. Αυτό το ειδικό σύστημα που υιοθετήσαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρείται αναφορά σύστημα πλέον παγκόσμια ιδιαίτερα σε αγορές ε, μεγάλων εμπορικών εταίρων. Υπάρχουν κάποια θέματα όμως τα οποία εκκρεμούν. Για κάποια προϊόντα υψηλής οικονομικής ε, αξίας υπάρχουν ε, δυστυχώς τρευλές πρακτικές χρήσεις τους και καταχρήσεις στην ονομασία τους και θα πρέπει να υπάρχει έλεγχος όχι μόνο στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και παγκόσμια. Αυτό περιλαμβάνεται και στη στρατηγική που υιοθετήσαμε το 2014 και περιλαμβάνεται επίσης και στους στόχους της στρατηγικής μας ε, που δημοσιεύθηκε στις 14 Οκτωβρίου. Ε, ξέρετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει τις διαπραγματεύσεις και στα πλαίσια του ΠΟΕ. Θέλουμε να υπάρξει προστασία αυτών των αγαθών ε, και σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο έχει υπάρξει κάλυψη προϊόντων όπως τα Πνευματώδη και ο ίνος. Είναι όμως αναπόφευκτο ότι στο τέλος η κατάληξη ε, θα εξαρτηθεί από το επίπεδο φιλοδοξίας το οποίο ε, θα καταλήξει η υπουργική διάσκεψη στο τέλος του μηνός των Ναϊρόμπι. Ταυτόχρονα μια βασική προτεραιότητα ε, της ε, προσπάθειάς μας στα πλαίσια των διμερών διαπραγματεύσεων παραμένει το συγκεκριμένο θέμα. Ε, τέλος, πριν δώσω το λόγο, θα έλεγα να πω ότι η στρατηγική μας που δημοσιεύτηκε στις 28 Οκτωβρίου λέγει ότι εμείς θα προσπαθήσουμε να χρησιμοποιήσουμε τις παραδοσιακές τεχνοτροπίες και να δούμε αν μπορούμε να διευρύνουμε την ονομασία αυτή και σε μη γεωργικά προϊόντα. Ευχαριστώ. Τζον Κλάρκ ονομάζομαι. Είμαι ε, αναπληρωτής ε, διευθυντής για τα ζητήματα γεωγραφικών ενδείξεων στην DG Agri της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ας θυμηθούμε όλοι λίγο τι είναι η γεωγραφική ένδειξη. Η γεωγραφική ένδειξη αποτελεί πνευματικό δικαίωμα το οποίο ισοδυναμεί με δίπλωμα βρεσιτεχνία ή με εμπορικό σήμα. Πρόκειται για ένα προϊόν ευρεσιτεχνία η εμπειρογνωμοσύνη, τεχνογνωσία και η φήμη του προϊόντος τελικά συνδέεται με τη συγκεκριμένη γεωγραφική αυτή περιοχή. Υπάρχει μια αιτιώδη συνάφεια, αν θέλετε, ανάμεσα στο προϊόν και στο χώρο παραγωγής του. Όπως είπε και ο συναδελφός μου, οι γεωγραφικέ ενδείξει έχουν πολύ σημαντική εμπορική αξία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ο μεγαλύτερο εισαγωγό ε, γεωργικών προϊόντων, αλλά και εξαγωγό ε, τροφίμων και γεωργικών προϊόντων, χάρη στις μεταρρυθμίσεις της ε, κοινή γεωργικής πολιτικής που κατάφεραν να κάνουν τον δικό μας τον κλάδο πιο ανταγωνιστικό. Έχουμε πλέον ένα πλεόνασμα στο εμπορικό ισοζύγιο του ε, αγροδιατροφικού τομέα, 17 δισεκατομμύρια περίπου ευρώ, και βλέπετε ότι οι γεωγραφικές ενδείξεις ουσιαστικά συμβάλλουν στις σημαντικότατες αυτές ε, οικονομικές επιδόσεις. Πέρυσι περίπου 15 δισεκατομμύρια ευρώ είναι οι εξαγωγές μας σε γεωγραφικές ενδείξεις και ακριβώς επειδή τα προϊόντα αυτά ουσιαστικά αντιστοιχούν στην ιδιαίτερα υψηλή ποιότητα των ευρωπαϊκών προϊόντων, μπορούμε να πούμε ότι τα προϊόντα γεωγραφικών ενδείξεων έχουν γενικότερα θετική επίπτωση και στα υπόλοιπα προϊόντα τα οποία εξάγουμε στον κόσμο. Τώρα, για ποιο λόγο οι γεωγραφικές ενδείξεις είναι τόσο σημαντικές για την αγροτική μας οικονομία, καθώς επίσης και για το εμπόριο, την οικονομία και την απασχόληση. Καταρχάς, οι γεωγραφικές ενδείξεις δεν αποτελούν προνόμιο δύο-τριών κρατών μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Από τότε που τη δεκαετία του 90 δημιουργήσαμε ένα ευρύτερο καθεστώ για τι γεωγραφικέ ενδείξει, όλο και περισσότερα κράτη-μέλη ενδιαφέρθηκαν για το σήμα τη γεωγραφική αυτή ένδειξη. Επομένω, όλα τα κράτη-μέλη πλέον προστατεύουν τι γεωγραφικέ του ενδείξει. Δεν μιλάμε μόνο για σαμπάνια, προσούτο τη Πάρμα ή σκοτσέζικο ουίσκι. Αναφερόμαστε επίση και σε λετωνικά, γερμανικά, σουηδικά προϊόντα, τα οποία καλύπτονται από γεωγραφική ένδειξη. Επίση, οι γεωγραφικές ενδείξεις προσδίδουν περισσότερη αξία. Δεν αφαιρόμαστε απλώς σε κάποια προϊόντα αυτή τη στιγμή, αλλά γενικότερα στην εξαγωγή προϊόντων υψηλής ποιοτικής αξίας που ζητάνε πάρα πολλοί πελάτες σε διάφορες ξένες αγορές. Χθε, για παράδειγμα, ο Υπουργός Γεωργίας των ΗΠΑ είπε ότι όντως υπάρχουν πάρα πολλοί πελάτες και στην Αμερική οι οποίοι προτίθενται να πληρώσουν περισσότερα χρήματα προκειμένου να έχουν ένα ευρωπαϊκό προϊόν το οποίο καλύπτεται από γεωγραφική ένδειξη και πολλές φορές η τιμή αυτή μπορεί να είναι και διπλάσια ενός προϊόντος που δεν έχει γεωγραφική ένδειξη. Βλέπουμε επίση πολλέ φορέ ότι οι γεωγραφικέ ενδείξει και τα σχετικά προϊόντα προκύπτουν κυρίω από μικρού παραγωγού, μικρού αγρότε και μικρομεσαίε επιχειρήσει που απασχολούν πάρα πολλού εργαζόμενου, Για παράδειγμα, όσοι εργάζονται για την παραγωγή παρμιτζάνο ρετζάνο στην Ιταλία είναι 50.000. 8.000 είναι τα άτομα που εργάζονται για την παραγωγή του τυριού κοντέ στη Γαλλία. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το μέσο αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για να αποφευχθεί η μετεγκατάσταση οποιασδήποτε παραγωγική δραστηριότητα σε άλλε περιοχέ εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, τι διαπραγματευόμαστε αυτή τη στιγμή. Καλύτερη προστασία και επιβολή της νομοθεσίας για τις γεωγραφικές ενδείξεις, σαν να είναι πνευματικά δικαιώματα δηλαδή. Όπως και τα πνευματικά δικαιώματα προβλέπεται η διαδικασία επί Να σας δώσω εδώ πέρα κάποια παραδείγματα. Τη φέτα για παράδειγμα, το οποίο παράγεται στην Αυστραλία, το οποίο παρουσιάζεται ως ελληνικό προϊόν, προσούτο το οποίο παρουσιάζεται ως Ιταλικό, ενώ δεν είναι, βλέπετε και την Ιταλική σημαία και βλέπετε εδώ πέρα ένα πακέτο με δαμάσκηνα από την Αζόν της Γαλλίας, τα οποία παράγονται στην Καλιφόρνια και πολλούνται στην Ιαπωνία. Καταλαβαίνετε ότι τα παραποιημένα αυτά προϊόντα ουσιαστικά προκαλούν πολύ μεγάλη ζημία και στους, και στους παραγωγούς και επίσης βάλουμε κατά της φήμη των προϊόντων απέναντι στους ε, καταναλωτές. Βλέπετε εδώ πέρα ότι χρησιμοποιούνται και κάποια άλλα «η ελαφίνα που πλήττει», bore dog, κατά λέξη η ελαφίνα που πλήττει, η goat ρωτή, παρουσιάζονται ως ε, κρασί ε, μπορντό για παράδειγμα. Καταλαβαίνετε ότι και πάλι εδώ πέρα η ζημία είναι πάρα πολύ σημαντική για τα προϊόντα αυτά και πάλι αυτή η πρακτική βάλει κατά της φήμη των προϊόντων τι προσπαθούμε εμεί τώρα να πετύχουμε στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων που έχουμε για τι γεωγραφικέ ενδείξει. Τέσσερα πράγματα. Πρώτον, υψηλό επίπεδο προστασία για τους εταίρους μας, για τις αγορές μας, τουλάχιστον όσον αφορά το άρθρο 32 TRIPS για τα τρόφιμα, Επίσης, διοικητική επιβολή από τις κυβερνήσεις των ανάλογων μέτρων, γιατί αν ένας παραγωγός μπορεί να επιβάλλει τα δικαιώματά του μόνο ένδικα μέσα από το δικαστικό σύστημα, καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι πάρα πολύ δαπανηρό. Και ξέρετε ότι η περισσότερη παραγωγή προϊόντων γεωγραφικών ενδείξεων είναι μικρή παραγωγή και δεν έχουν τα χρήματα για να προσφύγουν κατά ενό Κινέζικου, Καναδικού ή Αμερικανικού δικαστηρίου. Επίση, προσπαθούμε να έχουμε μια συνύπαρξη ανάμεσα στα υφιστάμενα GIs και τα προηγούμενα εμπορικά σήματα τα οποία ισχύουν και στην Ευρώπη αλλά και σε πολλές άλλες χώρες. Και αυτό προβλέπεται πάλι στη Συμφωνία TRIPS. Και τέταρτον, στις διάφορες συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών έχουμε έναν κατάλογο προστατευμένων προϊόντων βιογραφικών ενδείξεων. Η ίδια δηλαδή η συμφωνία περιλαμβάνει τη δέσμευση προστασίας και επιβολής νομοθεσίας όσον αφορά τα προϊόντα γεωγραφικών ενδείξεων. Όπω είπε ο αδελφό μου, σε πολυμερέ επίση επίπεδο, στα πλαίσια του ΠΟΕ προσπαθούμε να προασπίσουμε τι γεωγραφικέ ενδείξει στα πλαίσια του, της αναπτυξιακής ατζέντα του Ντόχα. Δυστυχώ όμω δεν έχουμε καταφέρει να πετύχουμε πρόοδο και δεν νομίζουμε ότι θα επιτευχθεί πρόοδο στη σύνοδο του Ναϊρόμπι. Επίση, στα πλαίσια του WIPO, του Παγκόσμιου Οργανισμού προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας προσπαθούμε να πετύχουμε μία συμφωνία μέσω της οποίας τα κράτη-μέλη θα μπορούν και σε διμερές επίπεδο να προστατεύουν τα προϊόντα γεωγραφικών ενδείξεων. Όπως καταλαβαίνετε όμως επικεντρωνόμαστε πάρα πολύ στις ε, διμερείς ε, σχέσεις που έχουμε. Βλέπετε εδώ πέρα στο χάρτη αυτό καταρχάς ποιες είναι οι χώρες με τις οποίες έχουμε συμφωνίες όσον αφορά τον ίνο και τα ενοπνευματόδη. Βλέπουμε έπειτα και τις χώρες εκείνες όπου έχουμε μια ευρύτερη συμφωνία στα πλαίσια ε, ε, συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών, Καναδάς, Κορία κτλ. Και έχουμε βέβαια και τις διαπραγματεύσεις οι οποίες ολοκληρώθηκαν πρόσφατα με το Βιετνάμ, όπου έχουμε προστασία 150 περίπου ονομασιών. Και έχουμε βέβαια και τη διαδικασία με την Ιαπωνία, η οποία είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα αγορά, όχι μόνο για το σκοτσέζικο ουίσκι, αλλά και για πολλά άλλα προϊόντα. Η Κίνα επίση είναι τεράστια αγορά για τα προϊόντα γεωγραφικών ενδείξεων τη Ευρώπη, όπου έχουμε πολλέ παραποίησει. Έχουμε την Ινδία, το Μερκοσούρ, αλλά προσπαθούμε να πετύχουμε και προστασία 250 εισαγόμενων προϊόντων γεωγραφικών ενδείξεων στα πλαίσια της TTIP, συμφωνίας με, τον, με τις Περισσότερα στοιχεία μπορείτε να δείτε και στην ανακοίνωσή μας. Περιλαμβάνουμε επίσης την ε, Αυστραλία, τη Χιλή και το Μεξικό. Πάντως ε, Όσον αφορά την συμφωνία TTIP, είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε στη συμφωνία αυτή να διασφαλίσουμε αυτά τα προϊόντα, τα οποία διασφαλίζονται εκεί πολύ περισσότερο από ό,τι στι υπόλοιπε συμφωνίε ελεύθερων συναλλαγών. Ξέρουμε ότι οι διαπραγματεύσει είναι δύσκολε αυτή τη στιγμή στα πλαίσια τη TTIP. Με τη συνεργασία των ΗΠΑ θέλουμε να προστατεύσουμε όχι μόνο τα γεωργικά μα προϊόντα και τα τρόφιμα, αλλά να αποφύγουμε και οποιασδήποτε δικαστικές διαφορές οι οποίες είναι ιδιαίτερα δαπανηρές καθότι πρέπει να προσφύγουμε στα αμερικανικά δικαστήρια. Θέλουμε επίσης να αποφύγουμε σήματα εθνικά τα οποία θα μπορούσαν να μην ενημερώσουν σωστά τον καταναλωτή και να τον παραπλανήσουν, σημαίε για παράδειγμα κτλ. Και προσπαθούμε επίση να βρούμε συγκεκριμένε λύσει όσον αφορά κοινόχρηστε ονομασίες κάποιων προϊόντων. Δεν ζητάμε όμω στα πλαίσια τη TTIP να μεταρρυθμίσει το σύστημα πνευματικών δικαιωμάτων οι Ηνωμένε Πολιτείε, ούτε προσπαθούμε στα πλαίσια της TTIP να ανακαλέσουμε ή να μονοπολίσουμε κάποια ονόματα τα οποία θεωρούνται γενικά τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θέλουμε απλώς να φαίνεται ξεκάθαρα μέσω αποδεικτικών στοιχείων αυτό. Επίσης και σε αντίθεση με αυτό που είπαν ορισμένοι Αμερικανοί, δεν προσπαθούμε να προασπίσουμε απλά ευρωπαϊκά ονόματα, προσπαθούμε απλώς να προασπίσουμε όντως προϊόντα τα οποία φέρνουν γεωγραφική ένδειξη. Δεν προσπαθούμε να καλύψουμε ονομασίες όπως προβολόνε, μοτσαρέλα, πίτσα τσίζα ε, κτλ. Δεν θα έπρεπε λοιπόν να πιστεύετε τους Αμερικανούς συνομιλητές που λένε κάτι τέτοιο. Στα πλαίσια διαπραγματεύσεων αυτών οι Ηνωμένε Πολιτείε, μολονότι είχαν αρχικά κάποιε ενστάσει στο να βρουν μία λύση για τι γραφικέ ενδείξει, στι δικέ του συμφωνίε ελεύθερων σταλεγών φροντίσουν να προστατεύσουν τα δικά του αμερικανικά προϊόντα, τι αμερικανικέ γεωγραφικέ ενδείξει. Και στα πλαίσια τη TTIP, οι Αμερικανοί, προστατεύουν το whisky το το bourbon, δεν αποκαλούν τα προϊόντα τους προϊόντα γεωγραφικών ενδείξεων, αλλά ουσιαστικά καταλήγουν στο ίδιο αποτέλεσμα. Καταφέρνουν τελικά να προστατεύσουν στις συμφωνίες τέτοιων Σταλλαγών προϊόντα γεωγραφικών ενδείξεων. Επίσης, όσον αφορά την TTIP, είναι ιδιαίτερα θετικό ότι οι ΗΠΑ δέχθηκαν ότι οι γεωγραφικές ενδείξεις θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο ανάλυσης στα πλαίσια του TTIP, που θα πρέπει να ενταχθούν σε αυτή τη συμφωνία και βέβαια έχει επιμείνει ιδιαίτερα γι' αυτό και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ξέρετε ότι είμαστε λιγότερο ανταγωνιστικοί στον τομέα τη γεωργία σε σχέση με τι ΗΠΑ. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε εμεί κάποιε παραχωρήσει στον τομέα αυτό στα πλαίσια του TTIP και είναι πολύ σημαντικό να καταφέρουμε, διασφαλίσοντα γεωγραφικές ενδείξει να προστατεύσουμε ισορροπημένα του δικού μα του παραγωγού. Αυτή τη στιγμή είναι αντιτιθέμενε οι απόψει ε, Ευρωπαίων και Αμερικανών. Η Αμερικανική πλευρά θεωρεί ότι δεν μπορεί να δεχθεί εύκολα τα δικά μα αιτήματα. Από την άλλη όμω, προτείνει να μειώσουμε το δικό μα επίπεδο προστασία στην Ευρώπη, να αποδυναμώσουμε δηλαδή το δικό μα ε, σύστημα IPR, προκειμένου Αμερικανική παρμεζάνη, Αμερικανική φέτα... Να... δεν πρόκειται πολύ απλά να συμβεί. Και καταλαβαίνετε ότι και εμείς επιμένουμε στο να μην χρησιμοποιούνται από την αμερικανική πλευρά κάποιοι όροι όπως κιάντι, σαμπάνια κτλ. Πρέπει λοιπόν να σημειωθεί ακόμα σημαντική πρόοδος όσον αφορά την προστασία των προϊόντων γεωγραφικών ενδείξεων στα πλαίσια του TTIP. Σίγουρα θα έχουμε δυσκολίες αλλά προσβλέπουμε και στην υποστήριξη της δικής σας της ε, Επιτροπής. Η συμφωνία αυτή για τις γεωγραφικές ενδείξεις θα είναι πάρα πολύ σημαντική και αποτελεί ένα απόσπαστο τμήμα μιας μελλοντικής συμφωνίας TTIP. Σας ευχαριστώ πολύ. ευχαριστώ πολύ κύριε Κλάρκ. Μας έδωσαν 10 λεπτά παραπάνω οι διερμηνείς. Όμω αυτά τα 10 λεπτά πέρασαν και θα συνεχίσουμε στα αγγλικά. Ευχαριστούμε λοιπόν του διερμηνείς για τα 10 λεπτά και τώρα συνεχίζουμε την συζήτηση στα αγγλικά. Begin and Madame e Finish the interpretation.